Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε Βίλμπαξ, αξιότιμοι φιλοξενούμενοι. Εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση αυτή που έχουμε σήμερα με θέμα ανάπτυξη και εκπαίδευση. Ονομάζομαι Φίλιπ Κασμάρη, είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής Ανάπτυξης και είναι ιδιαίτερα τιμή για μένα που φιλοξενώ εδώ εσάς και τον Επίτροπο Πίλπαξ. Ελπίζω ότι θα περάσουμε καλά σήμερα. Έχουμε δύο πάνελ. Το πρώτο πάνελ αναφέρεται στην ανάπτυξη και στην ε, ανάπτυξη και την εκπαίδευση και το δεύτερο πάνελ έχει να κάνει με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση. 20 λεπτά θα αφιερώσουμε μετά από κάθε πάνελ για την ανταλλαγή απόψεων, σχόλια από τους συμμετέχοντες, ε, τους ευρωβουλευτές κλπ. Επιτρέψτε μου επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει, συνδέεται άμεσα με μια έκθεση φωτογραφίας που έχουμε όσον αφορά την ανάπτυξη και την εκπαίδευση, έτσι όπως το είδαν φωτογράφοι Πολωνοί. Είναι στα πλαίσια της Πολωνικής ε, Προεδρίας. Ο κύριος ε, Στενέσκη, υφυπουργό για την Ανάπτυξη στην Πολωνία, είναι επίσης εδώ μαζί μας. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι να συμμετάσχετε στα γένεια της ε, έκθεσης αυτής φωτογραφίας που θα λάβουν χώρα σήμερα στις 6.30 στον τρίτο όροφο, στο Space Bar όπως ονομάζεται. Επίσης θέλω να καλωσορίσω θερμά εδώ τον Επίτροπο Μπίλβαξ, ο οποίος θα κάνει κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση, τη συνειδητοποίηση του κόσμου για το θέμα αυτό κλπ. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, η διαβούλευση που γίνεται με όλους τους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας διαρθρωμένου διαλόγου, η οποία μας επιτρέπει να μάθουμε την άποψη όλων των εταίρων ανά τον κόσμο, τη γνώμη τους, τι έχουν να προτείνουν όσον αφορά το θέμα αυτό. Και η δεύτερη πρωτοβουλία είναι μελέτη που γίνεται στην Ευρώπη για ανάλυση όσον αφορά την αναπτυξιακή παιδεία με εμπειρίες από την Ευρώπη και με συστάσεις. Δίχως άλλο θα ακούσουμε πολύ περισσότερα για τη δουλειά αυτή κατά τη διάρκεια του πρωινού. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ τον Επίτροπο Πιλ Βάλξ, ο οποίος πολύ συχνά έρχεται στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αξιότιμοι επισκέπτες κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ανέλαβαν να οργανώσουν την ακρόαση αυτή. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολούνται με το θέμα αυτό, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. Πρέπει να ξέρετε ότι τον προηγούμενο Οκτώβριο είχαμε και εμείς μια τέτοια διάσκεψη και τώρα πολύ χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσά εδώ. Ήμουνα δάσκαλος, διευθυντή σχολείου και πάντα με ενδιαφέρε πάρα πολύ το θέμα της εκπαίδευση. Και όσο περνάει ο καιρός με ενδιαφέρει όλο και περισσότερο. Και όσο περνάνε τα χρόνια και προχωράω στην καριέρα μου, ε, πιστεύω όλο και περισσότερο στην δύναμη που έχει η αναπτυξιακή παιδεία. Και όλο και περισσότερο πιστεύω ότι η ανάπτυξη είναι κάτι πολύ δυνατό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ήμουν επίτροπο για την ανάπτυξη κάποια στιγμή και πιστεύω ότι η αναπτυξιακή παιδεία εξακολουθεί να έχει τεράστια σημασία. Γιατί πρόκειται για τη συνειδητοποίηση του κόσμου έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση μέσα στην οποία το ευρωπαϊκό κοινό ενδιαφέρεται για τα αναπτυξιακά θέματα και είναι Έτοιμο ο κόσμος να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Και τη συνειδητοποίηση αυτή του κόσμου τη χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή του. Όχι μόνο για να στηρίξουμε την αναπτυξιακή μα πολιτική και τους στόχους της, αλλά πάνω απ' όλα για να δημιουργήσουμε το μέλλον τη Ευρώπης, να του δώσουμε σάρκα και οστά. Κάτι πολύ σημαντικό σήμερα για όλου. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ε, τη σημασία και τα θετικά της αναπτυξιακής ε, παιδείας. Τα γνωρίζετε όλα πολύ καλά. Κατά τη γνώμη μου αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να χτίσουμε πάνω στις μέχρι τώρα επιτυχία μας και πώς θα καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα. Από πλευράς λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας το πρόγραμμα DEAR για παράδειγμα, έτσι ώστε καταλητικά να βοηθήσει τα διάφορα προγράμματα τα οποία ήδη λαμβάνουν χώρα στις χώρες μέλη και να ενισχυθούν τέτοια προγράμματα σε όλες τις χώρες μέλη. Έτσι λοιπόν η αναπτυξιακή παιδεία ε, γι' αυτό αποτελεί και προτεραιότητα. Η αναπτυξιακή παιδεία για παράδειγμα στα σχολεία. Αν οι αυριανοί Ευρωπαίοι θέλουμε να μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο έτσι ώστε να δώσουν μορφή στο μέλλον, πρέπει να τους βοηθήσουμε ώστε να νιώθουν ε, πολίτες του κόσμου. Οι συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-μέλη για σχετικά με την αλληλεγγύη σε έναν μελλοντικό κόσμο είναι κάτι πολύ βασικό και για μας. Επίσης χαίρομαι πολύ που διαπιστώνω ότι πολλές χώρες μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τσεχία πιο πρόσφατα για παράδειγμα έχουν υιοθετήσει στρατηγική για την αναπτυξιακή παιδεία. Τέτοιες στρατηγικές στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν καρπό μιας ε, μακράς διαδικασίας όπου συμμετέχουν όλοι σε εθνικό επίπεδο και δείχνουν πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος στην Ευρώπη για την αναπτυξιακή παιδεία. Στη χώρα μου, την Λετωνία, έχουμε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται School, σχολεία, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στόχος είναι να καταρτήσουμε τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς για την αναπτυξιακή παιδεία και αποτελεί μια βάση για την ε, παρετέρω δουλειά μας. Πρωτοστατεί το Υπουργείο Παιδείας στην αναπτυξιακή αυτή παιδεία ε, καταρτίζοντας τους διδάσκοντες πρώτα απ' όλα, αλλά και άλλες χώρες, και η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. έχουν τέτοιες στρατηγικές για ε, συνδυτοποίηση των διδασκόντων πρώτα απ' όλα. Και δημιουργούνται επίσης και σχέσεις πιο στενές ανάμεσα στους ε, ε, διδάσκοντες, τους μαθητές και τους ομολόγους τους από την άλλη πλευρά, στο Αφγανιστάν για παράδειγμα. Έτσι θα πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι στόχοι για τους ανθρώπους σε, στις υπονάπτυξη χώρες. Τι σημαίνει για το μέλλον τους, τι σημαίνει για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάπτυξης στην πράξη και πώς τα αντιμετωπίζουν. Θα μπορούσα να σας δώσω και άλλα παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα λίγα δίνουν μια εικόνα του τι μπορούμε να κάνουμε παρετέρω έτσι ώστε η αναπτυξιακή παιδεία να εξακολουθήσει να είναι ζωντανή και να περάσει στα χέρια της επόμενης γενιάς. Φυσικά η δουλειά μας για την αναπτυξιακή παιδεία δεν πρέπει να σταματάει στις πόρτες των σχολιών. Όχι. Χρειάζεται συνειδητοποίηση μεταξύ όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτή είναι εξίσου σημαντική. Και γι' αυτό και χρώμαστε πάρα πολύ για διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τους ενήλικες. Με εκστρατείες για συνειδητοποίηση του κόσμου σχετικά με διάφορα θέματα, όπως είναι η παγκόσμια δικαιοσύνη, το σωστό εμπόριο, το ηθικό εμπόριο, στόχοι της χιλιετίας. Πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία σε αυτή τη διαδικασία αποδίδει καρπούς. Και αυτό είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεχίσει αυτή την ειδική σχέση που έχει ήδη ξεκινήσει με όλους τους ε, εταίρους μας. Είμαι πεπισμένος ότι αποτελεί πρόσθετη αξία η συνεργασία μας αυτή με όλους τους εταίρους, με όλους όσους δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Έχουμε την περίοδο 2014-2020. Εγώ πρότεινα να εξορθολογήσουμε τα θεματικά προγράμματα. Αν η πρότασή μου εγκριθεί, τότε θα οργανωθούν εκ νέου με νέα προγράμματα διάφορες δραστηριότητες με συμμετοχή των τοπικών αρχών και θα φροντίσουμε ε, να δούμε καλύτερα τους στόχους του κόσμου με θέματα όπως είναι το κλίμα, η επισητιστική ασφάλεια, ε, επένδυση στους ανθρώπους κλπ. κλπ. Πρότεινα επίσης να αυξήσουμε και τα προγράμματα, τα μη κρατικά, ε, κατά πολύ μέσα στην επόμενη αυτή περίοδο. Η συνειδητοποίηση του κόσμου πρέπει να αποτελεί μέρος τέτοιου προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λοιπόν προσπάθειες και σε άλλα μέτωπα για να αναπτύξει περισσότερο στρατηγικές αναπτυξιακής παιδείας. Η αναπτυξιακή παιδεία και συνειδητοποίηση του κόσμου είναι πρωτοβουλία που περιλαμβάνεται στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου που οργανώνουμε. Αυτή η διαδικασία με συμμετοχή όλων και συνεργασία βέβαια οδηγεί σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Έτσι ανανεώνουμε τα σημεία τα οποία υπογραμμίζουμε, διότι δίνουμε περισσότερη σημασία σε σαφή πλαίσια για την αναπτυξιακή μας παιδεία και για τις δράσεις μας. Όλα αυτά, μαζί με τα αποτελέσματα από τη μελέτη DIR, θα οδηγήσουν σε προτάσεις που θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Έτσι λοιπόν υπογραμμίζουμε όλο και περισσότερο την ευρωπαϊκή διάσταση στα διάφορα προγράμματά μας και την γεωγραφική ισορροπία αυτών. Θέλουμε να υπάρχει υποχρέωση συμπληρωματικότητας επίσης με τις ε, πολιτικές των κρατών μελών και των στρατηγικών που έχουμε για τα προγράμματα ε, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τέτοιου είδους προσεγγίσεις και προγράμματα θα καθοριστούν πιο ξεκάθαρα στο μέλλον. Θέλουμε επίσης να εισακάγουμε και τη δυνατότητα στήριξης μεγάλων προγραμμάτων που ε, αποδεικνύουν ότι έχουν μια πολύ ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση. Είμαι σίγουρος ότι η διαδικασία που ξεκίνησε με την μελέτη αυτή θα συνεχίσει να έχει επιπτώσει στη δουλειά μας μια που συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την δουλειά μας και τη συνεργασία μας. Γνωρίζω ότι αρκετοί συμμετέχουν ακόμα στην μελέτη DIR από εσά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το κάνετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να συνεχίσει τη δουλειά της και στο DIR και να συνεχίσει να συμμετέχει σε προγράμματα και θα λάβουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα των σημερινών πάνελ για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προδεύσουμε περισσότερο όσον αφορά την αναπτυξιακή παιδεία. Κυρίες και κύριοι, η αναπτυξιακή παιδεία δίνει καρπούς όταν συμμετέχουν πολλοί και βοηθούν την πρόθεσή της και νοιάζονται ώστε το γενικό κοινό και οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά μπορούν να ενσωματωθούν σε μια τέτοια παιδεία. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, αλλά και πολλοί που δεν βρίσκονται εδώ, ξέρουν ότι τα θέματα της ανάπτυξης πρέπει να περνάνε από τα παιδιά. Δεν ε, είναι κάτι που διαφέρει από τη δικιά μας την προσέγγιση. Πιστεύω πάντως ότι εμείς είμαστε στο σωστό δρόμο. Πρέπει να επιταχύνουμε βέβαια ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις δικές σας αντιδράσεις για το τι λειτουργεί καλά και για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα για να πετύχουμε περισσότερα. Σε αυτούς τους δύσκολους και περίπλοκους καιρούς που ζούμε και στην Ευρώπη αλλά και όχι μόνο, καταλαβαίνετε ότι οι νέοι ανησυχούν για το μέλλον τους. Ε, ανησυχούν για την χρηματοδότηση προγραμμάτων σε τρίτες χώρες. την... Ε, πιστεύω όμως ότι η αναπτυξιακή παιδεία, παρόλο που μπορεί να μην γίνεται πάντα αρκετά κατανοητή, είναι θεμελιώδης. Και πιστεύω ότι πρέπει γι' αυτό να κάνουμε ακόμα περισσότερες προσπάθειες ώστε να πετύχουμε όχι μόνο τη γενική στήριξη υπέρ της ανάπτυξης, αλλά μια πραγματική συμμετοχή των πολιτών μας αυτή. Πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα της αντιλήψης πρέπει να στηρίξουμε δράσεις και να αγωνιστούμε γι' αυτό. Και πρέπει πάνω απ' όλα να αναρωτηθούμε. Πετυχαίνουμε το στόχο μας. Ε, υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να κάνουμε. Η, τα μηνύματά μας περνάνε όντως στο κοινό. Επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών μας. Όλοι μαζί πρέπει να πάρουμε αυτό το δρόμο και να υποβάλουμε αυτές τις ερωτήσεις στους εαυτούς μας. Η αναπτυξιακή παιδεία αξίζει τον κόπο. Έχει νόημα. Είναι μια από τις λίγες δραστηριότητες που τις νιώθει ο κόσμος στην Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας από τους κύριους δωρητές για την αναπτυξιακή παιδεία. Είμαι πεπισμένος ότι τα 31 εκατομμύρια ευρώ που κατά μέσο όρο δίνονται ε, κάθε χρόνο για το πρόγραμμα DEAR είναι χρήματα που πιάνουν τόπο. Ορισμένοι μπορεί να πούν ότι θα έπρεπε κατευθείαν να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εγώ όμως έχω να πω ότι αυτό ακριβώς κάνουμε. Επενδύουμε για την αναπτυξιακή παιδεία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι βλέπουμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα και επενδύουμε στον κόσμο παντού επενδύουμε στον κόσμο, ήδη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα παιδιά, στους ενήλικες, που ενδιαφέρονται και ξέρουν ότι μπορούν να βοηθήσουν και ότι θα έχουν κέρδος από αυτό, γιατί είναι πολίτες του κόσμου. Και μέσω των δραστηριοτήτων τους, μέσω της συμμετοχής τους, ξέρουν ότι με τη σειρά τους θα επενδύσουν περισσότερο πάνω στον κόσμο. Γιατί είμαστε μέσα σε ένα κόσμο που αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα. Δεν είναι ευγενή αυτό ο στόχο. Αν δεν είναι αυτό ευγενή στόχο, τότε ποιο είναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Και ο Διευθυντή Κρίστερσεν πρέπει να ξέρετε ότι είναι εδώ και ότι εκείνο είναι στη διάθεσή σα για να απαντήσει σε ό,τι ερωτήσει τεθούν όσον αφορά τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί ναι, δίνουμε μεγάλη σημασία στην αναπτυξιακή παιδεία και πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα που είχαμε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Commissioner, for your... Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και για τον λόγο και για την εμπλοκή σας στο θέμα. Ε, απαντήσετε στο γιατί χρειάζεται η αναπτυξιακή παιδεία. Ήδη δηλαδή τον τίτλο του πάνελ μας και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να συζητούμε το θέμα αυτό. Η αναπτυξιακή παιδεία είναι ευρεία έννοια που μπορεί να συμπεριλάβει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Κάποια τα αναφέρεται. Αύξηση της επίγνωσης, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, ε, υποστήριξη, εκστρατεία, μια συγκεκριμένη δράση με τίτλο Global Education, με την αναπτυξιακή παιδεία δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι για μας, έχει ήδη ξεκινήσει στην Πολωνία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πάνω από 10.000 μαθητές που παρακολούθησαν ένα μάθημα για την παγκόσμια εκπαίδευση στην περιφέρειά μου και μόνο. Άρα μπορούμε να επηρεάσουμε για τα σχολεία. Εδώ θα εξετάσουμε τις διάφορες προσεγγίσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη για να υπάρξει μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπτυξιακή παιδεία και γι' αυτό καλέσαμε εκπροσώπους από το Σύμβουλο της Ευρώπης, την Κοινωνία των Πολιτών, τα κράτη-μέλη και τον ακαδημαϊκό χώρο για να μας παρουσιάσουν διαφορετικέ προοπτικές και να ανοίξουν μια ευρεία συζήτηση με τους συμμετέχοντες στην ακρόαση. Θέλω να καλωσορίσω του πρώτου τρει ομιλητέ μα σε αυτό το πρώτο πάνελ την κυρία Ντεώτη από το Πανεπιστήμιο του Όλου στη Φιλανδία, την Σουζάνα Γκλαβίτσκοβα, Διευθύντρια Αναπτυξιακή συνεργασία και Ανθρωπιστική βοήθεια στο, τμήμα, στο δύσκολο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών τη Τσεχία και τον Μάτια Φίτλερ, Διευθυντή του, της ε, Ιρλανδικής Εταιρείας Ανάπτυξης και ε, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου. Η κυρία Ανδρεώτη θα μιλήσει πρώτη για 8 λεπτά για να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Παρακαλώ. Is it okay now? Okay, thank you. So, ladies and gentlemen, uh... Κυρίες και κύριοι, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου που μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχω. Ήμουν δασκάλα από τη Βραζιλία. Ήμουν μετανάστης, μητέρα Ευρωπαίων πολιτών και γι' αυτό θεωρώ ότι η αναπτυξιακή παιδεία είναι κεντρικό στην δική μου προσωπική ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε, είμαι η μόνη διδάσκουσα στην Ευρώπη για την παγκόσμια εκπαίδευση. Ένα θέμα που νομίζω δημιουργεί μεγάλη ευθύνη. Θα παραπέμπω σε στοιχεία που δεν περιλαμβάνει το ενημερωτικό μου κείμενο. Καλό, αλλά, καλό λοιπόν να τα δείτε και αυτά. Μετά την τις επιθέσεις στο Όσλο και τις εξεγέρσεις στην Αγγλία είναι ακόμα σημαντικότερο να ε, μπορεί η παγκόσμια εκπαίδευση να επιτρέψει στους ανθρώπους να δράσουν με νέο τρόπο σαν παγκόσμιοι πολιτές σε ένα σύνθετο, άδικο, αβέβαιο ε, και άνισο κόσμο παρέχοντας ε, δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε την απογοήτευση και την, ε, από την πολιτική διαδικασία και την αύξηση της βίας. Η αναπτυξιακή παιδεία λοιπόν είναι κεντρική στην ανάπτυξη του ανθρώπου σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας ελεξάρτησης και ασφάλειας. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης, η αναπτυξιακή παιδεία πρέπει να αναγνωρίσει το, την αλλαγή του προφίλ των διδασκομένων, της διδαχής, της γνώσης, αλλά και των ίδιων των κοινωνιών και να προσφέρει παράλληλα τις ενδεδειγμένες παιδαγωγικές υποστηρίξεις που θα επιτρέψουν να έχουμε μια παγκόσμια εικόνα μέσω της κρίσης και να μπορούμε να λάβουμε υπόψη την πολλαπλότητα των απόψεων και να, δείξουμε την δυνατότητα να εμπλακούμε με πιο σύνθετο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τρεις διαστάσεις. Πρώτον, τη διάσταση της εναρμόνισης των πολιτικών ανάπτυξης στην αναπτυξιακής παιδείας στην Ευρώπη, δεύτερον την, ανά, την ανάγκη ε, δέσμευση, ισχυρή δέσμευση στην δεοντολογική και ε, ανάπτυξη και την ενίσχυση της υποστήριξης της εκπαίδευσης των δασκόνων. Για το πρώτο θέμα, την εναρμόνιση των πολιτικών ε, αναπτυξιακής παιδείας πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την μέχρι τώρα επιτυχία. Είχαμε επιτυχημένα προγράμματα χρηματοδοτημένα από την Επιτροπή σε πολλές χώρες. Στην Πορτογαλία, στην Τσεχία, την Πολωνία και τη Φιλανδία έχουμε μια σειρά πολιτικών που πραγματικά έχουν μια προβολή προς το μέλλον. Επίσης χρειάζεται ένας διάλογος, συνεχιζόμενος διάλογος και αμφίδρομος διάλογες. Θέλουμε η συνένεση να λειτουργεί σε μόνιμη βάση, να μην κλείνουμε τη δυνατότητα για περαιτέρω αλλαγέ σε περίπτωση αλλαγή του πλαισίου. Επίση, είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε πολλά παραδείγματα, πολλά υποδείγματα ανάπτυξη και θα τα αναφέρω στο τέλο τη παρουσίασή μου. Επίση, χρειάζεται να γνωρίσουμε τις διαφορετικέ αντιλήψει που υπάρχουν για την αναπτυξιακή παιδεία σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ε, υπάρχει μια έκθεση που λέγεται D-Watch Report η οποία είναι διαθέσιμη στην πρώτη σειρά εδώ που περιλαμβάνει μια σειρά ορισμών της αναπτυξιακής παιδείας ε, παγκόσμια εκπαίδευση, αύξηση της επίγνωσης η έκθεση αναφέρει λιτά ότι οι δημόσιες σχέσεις δεν είναι παιδεία, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε για να καταλάβετε λοιπόν το δικό μου πλαίσιο προέλευσης. Εγώ θεωρώ ότι η εκπαίδευση αυτή λειτουργεί ως, διαμε... ως κρίκο σύνδεσης μεταξύ του εγώ και του υπόλοιπου κόσμου με δυνατότητα ανάπτυξης και κατανόησης στο πλαίσιο της ευρύτερης ε, εκπαιδευτικής πολιτικής. Και που επιτρέπει να καταλάβουμε την παγκόσμια, τον παγκόσμιο καπιταλισμό, τις διεθνής μεταναστευτικές ζωές και την αναμόρφωση της πολιτικής ηγεσία. Η παγκόσμια λοιπόν εκπαίδευση και η αναπτυξιακή παιδεία είναι στο κέντρο αυτών των αλλαγών στην εκπαίδευση. Το ίδιο συνδέεται με τις διαφορές της τάσης εκπαίδευσης που εμφανίστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν στην εκπαίδευση εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα, τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ανάπτυξη και που συνδέουν την εκπαίδευση με το παγκόσμιο πλαίσιο. Η πολιτισμική εκπαίδευση, η ηθική εκπαίδευση περί της η δημιουργία της εικόνας του παγκόσμιου πολίτη είναι βασικά κομμάτια της, της εκπαίδευσης αυτής. Τώρα, τι δεξιότητες, τι προσόντα χρειάζονται για τους τρεις αυτούς κύκλους. Εγώ δούλεψα με, το, με την έννοια της παγκόσμιας νόησης. Μέσα σε ένα ε, υπάρχει μια δομή στην Φιλανδία που επιτρέπει την κινητικότητα και συνεργαστήκαμε. Η ιδέα λοιπόν αυτής της ε, παγκόσμιας νόησης είναι μία σειρά προσόντων και δεξιοτήτων που είναι σημαντική για να μπορέσουν οι διδασκόμενοι να έχουν μία πλήρη εικόνα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και της διαφορετικότητας της παιδείας με αύξηση της επίγνωση για τις παγκόσμιες διεργασίες για καλύτερη εικόνα των, για καλύτερη δυνατότητα αντιμετώπισης της, της παγκόσμιας και που θα περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα, την ικανότητα να, να, ανταποκριθεί στις, απα, στις απαιτήσεις, ευελιξία, ε, ανοιχτό μυαλό, με, συλλογιστική και αντιδραστική. Στα πλαίσια της αύξησης αυτής της επίγνωσης, ε, η ανοιχτή προσέγγιση, η αντιμε... ο σεβασμός του δικαιώματος των άλλων που έχουν αντίθετες απαντήσεις, αντίθετες απόψεις, η αμφισβήτηση όλων των δεδομένων είναι βασικά κομμάτια της εκπαίδευσης αυτής. Στο ίδιο πλαίσιο, η γνώση της ανισότητας, η πολυσυμμετοχή των πολιτών, η προσωπική εμπλοκή, η αντιμετώπιση και η άρνηση της ανισότητας, οι υπεύθυνε επιλογές είναι εξίσου βασικές παράμετροι. Σε ό,τι αφορά την ποικιλομορφία και την ανισότητα, θα ήθελα να σας καλέσω να δουλέψετε μαζί μου για να καταλάβετε κάτι που δεν συζητούμε συχνά. Μια διαδικασία που συχνά κάνουμε με φοιτητέ. Τους λέω, σκεφτείτε ένα λιβάδι με καλαμπόκια θερίζετε τα καλαμπόκια που τα βάζετε μπροστά σας. Έτσι μοιάζουν αυτά που μαζέψετε. Αυτό, αυτά είναι τα καλαμπόκια στην Νότια Αμερική, αλλά στην Ευρώπη βλέπετε ότι δεν μοιάζουν. Θα σου πούει ο κόσμος ότι αυτά τα καλαμπόκια δεν μοιάζουν με τα καλαμπόκια που βλέπουμε εμείς στο σούπερ μάρκετ. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην παγκόσμια εκπαίδευση πρώτα-πρώτα το θέμα της ηγεμονίας και του εθνοκεντρισμού. Κάτι που συνδέει την αναπτυξιακή παιδεία με την πολυπολιτισμική παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρότεινα να δοθεί έμφαση σε μια παγκόσμια ηθική πέραν των πατερναλιστικών και εθνοκεντρικών προσεγγίσεων να δοθεί έμφαση στην αμοιβαιότητα και την ε, αμοιβαία κατανόηση, να προχωρήσουμε από την ε, αλληλεξάρτηση για αγωιστικούς λόγους προς μια χρήση της ανάπτυξης ως μέσο για την αναγνώριση της αξιοπρέπειας ε, του ανθρώπου. Η παιδεία, η αναπτυξιακή παιδεία στο Νότο. Προτείνω να δώσουμε και εδώ έμφαση να τονίσουμε την ανάγκη για μεγαλύτερο διάλογο, εταιρική σχέση και συντονισμό. Στο πλαίσιο αυτό θα παραθέσω τον καθηγητή Χάρντιν Καρούμπα από το του Cape Town που ρώτησε η συνεργασία είναι μόνο συνεργασία μεταξύ θεσμών ή θέλουμε να υπάρχει ένας διάλογος, μία εμπλοκή που θα δημιουργεί πραγματική νέα γνώση και συνεργασία σε ό,τι αφορά τώρα την εκπαίδευση των διδασκόντων. Θέλω να παραθέσω το παράδειγμα της Φινλανδίας. Αυτό είναι ένα μάθημα που συντονίζω εγώ στο Όλου για την εκπαίδευση ε, των διδασκόντων σε θέματα ανάπτυξης, αναπτυξιακής παιδείας με έμφαση η ύλη στηρίζεται στην παγκόσμια νόηση, την ε, έμφαση στην ηθική, την επικεντρώνεται σε κοινωνικο-ιστορική παγκόσμια ανάλυση, ε, σχέση βορρά-νότου, ανατολή-δύση, την παγκοσμιοποίηση εκ των άνω και εκ των κάτω, κοινωνικά κινήματα, γεγονότα όπως το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα νέο παιδαγωγικό DNA του 21ου αιώνα με προσόντα που θα έχει στόχο όχι μόνο τη μεταβίβαση των πληροφοριών αλλά την ε, τις ηθικές επιλογές, τον εξοπλισμό, τον, την, την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να συμβιώνουν, δίνουμε έμφαση στην κινητικότητα, τη διεθνοποίηση και δίνουμε έμφαση σε μια ε, εκπαίδευση βάση της έρευνας. Εξού και η σημασία των ε, εμπειρικών μεθοδολογικών εργαλείων. Είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη και μεγαλύτερη έρευνα στον τομέα. Επίσης, το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δια εταιρικέ σχέσεις που περιλαμβάνουν εμπλοκή όχι μόνο διδασκόντων και διδασκομένων αλλά και της ευρύτερη κοινωνίας. Αυτά. Ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσω. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χαλαντίτσκοβα έχει το λόγο. morning. Καλημέρα σας. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω την στρατηγική ε, για την ε, αναπτυξιακή παιδεία στη χώρα μου διότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνησή μας και για το Υπουργείο Εξωτερικών τον οποίο, το οποίο είναι εκπροσωπό. Εγώ ε, προέρχομαι από το τμήμα της αναπτυξιακής ε, ε, παιδείας και βοηθείας και ε, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ε, διατυπώσουμε τη στρατηγική μας, ποιος ε, ανταποκρίνεται σε αυτήν τη διαδικασία και πώς προβλέπουμε να επιτύχουμε αυτή τη στρατηγική. Πρέπει να σας δώσω ορισμένα στοιχεία από την τσεχική δημοκρατία διότι αφού επανήλθαν στη δημοκρατία, προσπαθούμε ε, να συνδράμουμε στην επίλυση της ε, συνολικής ε, φτώχειας, αλλά θα πρέπει η προσπάθεια αυτή να στηρίζεται και από το κοινό και η συνειδητοποίηση του κοινού για τα θέματα αυτά ακόμη είναι σχετικά χαμηλή παρόλο που υπάρχει σαφής αλληλεγγύη των Τσέχων για τις ανθρωπιστικές κρίσεις, η ε, αναπτυξιακή βοήθεια και συνεργασία μακροπροθέσμως δεν είναι από τις πρώτες προτεραιότητες τους και δεν ε, φαίνεται να επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή. Για αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε όχι μόνο βάσει των δικών μας παρατηρήσεων αλλά συγχρόνως και βάσει των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των διαπιστώσεων τις οποίες έχουμε ε, κάνει να στηρίξουμε περισσότερο τις μη κυβερνητικέ μας οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο θέμα αυτό και αυτό μας οδήγησε στο να καταρτήσουμε μία εθνική στρατηγική η ε, στιγμή ήταν κατάλληλη διότι όταν ξεκινήσαμε πριν από δύο-τρία χρόνια μπορούσαμε συγχρόνως να ε, παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες ε, του Υπουργείου Παιδείας που παρακολουθούσε και ανέπτυσε το ε, σύστημα παιδείας της χώρας και από το 2003 βοηθάμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και υπάρχει γραμμή του προϋπολογισμού για μη κυβερνητικέ οργανώσεις που αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες και αποβλέπουν στην σύνδεση συνδρομή των δασκάλων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και της παιδείας και ε, έχουν συμβάλει στην προσπάθεια αυτή. Υπάρχει λοιπόν μία μικρή μεν συνδρομή η οποία όμως αναπτύσσεται όλο και περισσότερο κάθε επόμενο χρόνο ο φόρτος εργασίας τους δεν τους εμπόδισε να παρουσιάσουν πολλά στοιχεία και ε, να συμβάλλουν στην ε, στρατηγική. Ε, όλο και περισσότερες αρχές εκπαιδευτικές έχουν περιληφθεί στην στρατηγική. Υπάρχουν ε, διάφορα συνέδρια τα οποία έχουν αφιερωθεί στο θέμα αυτό για την ανάπτυξη της παιδείας όπως παραδείγματο χάρη το 2007 και ε, το 2008 στη χώρα μας. Ουσιαστικά η διαδικασία αυτή αποβλέπει ε, την διατύπωση ορισμένων στρατηγικών θεμάτων ε, στο να υπάρχει καλύτερο συντονισμός με τους βασικούς ε, εμπλεκομένους και να μπορέσουμε να δεχθούμε όσους ε, ε, προέρχονται από τον ε, χώρο της παιδείας αλλά και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία αυτά και από την ιστοσελίδα μας αλλά και από το έντυπο το οποίο έχουμε φέρει και μπορείτε να πάρετε όπου εμφανίζονται οι βασικές αρχές και οι βασικοί εμπλεκόμενοι καθώς επίσης και τα θέματα και, τα, και οι στόχοι τους οποίους έχουμε καταρτήσει για την επόμενη πενταετία. Χρησιμοποιούμε τον όρο global δηλαδή συνολικός, σφαιρικός κατά τρόπον ώστε να περιγράψουμε τα φαινόμενα τα οποία προσπαθούμε ε, να αντιμετωπίσουμε μέσω της στρατηγικής μας και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει να συμβιβαστούμε ε, με τις ε, απόψεις των εμπειρογνώμων από τη μία πλευρά και των αποδεκτών από τις άλλες και βλέπετε ότι προσπαθούμε να δούμε δούμε πόσο μπορεί ε, να επιληθούν τα διάφορα θέματα ε, που καθορίζει το Υπουργείο μας και πώς θα επηρεάσουμε και τους παράπλευρους τομείς ε, παραδείγματος χάρη παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις επιχειρήσεις για τον τρόπο της σκέψεως για πολυσχηδή παιδεία, όλα αυτά τα θέματα μας έχουν απασχολήσει. Και πρέπει να σας πω ότι γενικώ το θέμα είναι ε, προχωρά σωστά και υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση από τις ομάδες που συμμετέχουν στη διαδικασία καλύπτουμε τα διάφορα θέματα και προσπαθούμε ε, να μπορέσουν όλοι να αντιληφθούν ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων στις υποανάπτυξη και τις ε, ε, άλλες ε, χώρες διότι όπως είπα πρέπει όλοι να μπορέσουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ε, να υπάρχει άλλη λεξάρτηση, να καλύψουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα συνδυάσουμε με την αναπτυξιακή παιδεία. Θα είμαι σύντομη, αλλά όπως σας είπα, όλα τα θέματα αυτά ε, περιγράφονται ε, πιο εκτενώς ή στο έγγραφό μας. Καλύπτουμε και ορισμένες βασικές αρχές από την από την ε, ε, την ε, πλευρά ε, της δημοσίας παιδείας των μη κυβερνητικών οργανώσεων της επαγγελματική κατάρτασης της επιχειρησιακής συμμετοχής περιγράφονται επακριβώς τα καθήκοντα του κάθε κλάδου στο θέμα και καταλήγοντας θα ήθελα να σας πω ότι ο βασικός μας μας ε, στόχος είναι μέχρι το 2015 να έχουμε ε, τους στόχους αυτούς να περιλαμβάνονται στη διαβίου μάθηση και στο σφαιρικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως και ελπίζουμε ότι θα το επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ματίας Φίντλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως ο χρόνος περνάει, μου λέει 8 λεπτά, θα ξεκινήσω αμέσω, θα τα χρησιμοποιήσω όλα πιστεύω και ελπίζω να μην τα ξεπεράσω. Περνάω ευθύ αμέσω στο θέμα. Οι δύο προλαλήσαντες είπαν ότι η παγκόσμια εκπαίδευση, μάθηση, η αναπτυξιακή παιδεία είναι ένας πολύ καλός όρος για να εκφράσουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί πρόκειται εδώ πέρα για δύο τομείς, ε, δύο συζητήσεις, δύο ειδονιδές και πρόκειται για τις πολιτικές οι οποίες λαμβάνουν χώρο στα δύο αυτά θέματα. Η αναπτυξιακή παιδεία ξεκινάει με την συνεργασία ε, θυμόσαστε ότι είχαμε τους ιεραπόστολους, είχαμε διάφορους που πηγαίνουν και βοηθούσαν για την μόρφωση, για την ε, συνειδητοποίηση των ανθρώπων όσον αφορούσε τις εμπειρίες που είχαν ζήσει. Και έτσι σιγά σιγά προχωρήσαμε στην αναπτυξιακή παιδεία ενημερώνοντας τον κόσμο για το τι συμβαίνει στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία και οι στόχοι της χιλιετίας είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ανάπτυξη και με την εκπαίδευση. Πολλές συζητήσεις λοιπόν γίνονται και πολλές απαντήσεις πρέπει να δοθούν στον τομέα αυτό. Υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα για την γνώση, για τη μεθοδολογία με την οποία περνάει η γνώση. Όσοι όμως ασχολούνται με την αναπτυξιακή παιδεία πρέπει πολύ ξεκάθαρα να ξέρουν ποιε είναι οι συγκεκριμένες πολιτικές και να δουν πώς η αναπτυξιακή παιδεία θα περάσει στην διαδικασία μάθησης, στο curriculum, στο πρόγραμμα σπουδών. Πολύ βασικό θέμα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Βανέσα πριν τα ανέφερε όλα αυτά πολύ καλύτερα από ό,τι μπορώ να το κάνω εγώ για μένα. Το στοιχείο κλειδί εδώ είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή πώς ο κόσμος θα περάσει από την φιλανθρωπία στον σεβασμό. Πρέπει να βλέπουμε το θέμα της ε, ανάπτυξης από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δεν είναι το θέμα πώς ε, αυτοί που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά θα αναπτυχθούν για να φτάσουν στο δικό μας το μοντέλο. Όχι, υπάρχουν διαφορετικές ιστορίες. Και η αναπτυξιακή παιδεία αποτελεί ακριβώς μια πρόκληση προς αυτή την κατεύθυνση. Όσοι δουλεύουν στην αναπτυξιακή ε, παιδεία, ήδη από τη χώρα τους είναι πολύ συνδυτοποιημένοι. Έχουν δουλέψει πρώτα απ' όλα στις δικές τους της χώρας, έχουν ε, ασχοληθεί με θέματα παγκοσμιοποίησης και προσπαθούν να δουν πώς πράγματα τα οποία γίνονται σε τοπικό επίπεδο μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο παγκόσμιο επίπεδο. Ε, χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, δημιουργούν. Έπειτα, η διαδικασία μάθησης στην αναπτυξιακή παιδεία πρέπει να είναι συμμετοχική πρώτα απ' όλο, να συμμετέχουν πολλοί, να υπάρχει μεταφορά ε, γνώσης, πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της αλλαγής, να αλλάζουν τα πράγματα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αλλάξουμε τα πράγματα. Έπειτα υπάρχει το θέμα, όπως είπαμε, της συνδυτοποίησης, αλλά και το πώς θα νιώσει οι πολίτε του κόσμου κανείς. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να ενημερώνουμε ε, τους ανθρώπους μέσω της ανθρωπιστικής παιδείας για το τι συμβαίνει αλλού, αλλά πρέπει να τους κάνουμε να συνδυτοποιήσουν πώς μπορούν και εκείνοι να συμμετέχουν στις αλλαγές. Το θέμα δεν είναι να τους κάνουμε να σκεφτούν πω πω τη χάλι είναι ο κόσμος, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Όχι, το σημαντικό είναι να κάνουμε τον κόσμο να βρει τα μέσα και τον τρόπο να αλλάξει τα πράγματα. Υπάρχουν τέσσερα, τέσσερις διαστάσεις κλειδί κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι ο, οι αξίες και οι αντιλήψεις. Πολύ συχνά έχουμε την παραπληροφόρηση, έχουμε τις λάθος ιδέες, τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν σχετικά με την κατάσταση. Αξίες λοιπόν, πώς θα υπογραμμίσουμε τα θετικά, τις θετικές αξίες ε, του ανθρώπου και του πλανήτη. Πολύ βασικό. Τι αξίες είναι αυτές, πώς να νοιαζόμαστε για τους άλλους, πώς ε, να τους συμπονάμε, ε, πώς να νιώθουμε υπεύθυνοι. Για να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις αξίες χρειάζονται βέβαια ικανότητες, προσόντα, πρέπει κανείς να είναι λογικός, να μπορεί να επικοινωνεί με τον άλλον, ε, να τον καταλαβαίνει, να είναι επικριτικός. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε και πάνω στη γνώση με την αναπτυξιακή παιδεία. Δηλαδή δεν φτάνει απλώς να ξέρουμε αν ναι, εγώ μπορώ να κάνω αυτό. Όχι, πρέπει να γνωρίσεις καλά το αντικείμενό σου για να μπορέσεις να περάσεις τη γνώση της αναπτυξιακής παιδείας. Και η μάθηση γίνεται μέσω του κάνω. Μαθαίνω κάνοντας. Άρα χρειάζεται και στην πράξη να δουλεύει κανείς. Επειδή περνάει η ώρα και θέλω να σας μιλήσω για πολλά, θα συνοψίσω λίγο. Η ανάπτυξη, η αναπτυξιακή παιδεία, τι χρειάζεται. Χρειάζεται τη βοήθεια του κράτους, χρειάζεται μια παγκόσμια κοινωνία και χρειάζεται και ε, παραδείγματα γιατί χρειαζόμαστε τη συμμετοχή την κρατική. Ακούσαμε και πριν ότι χρειάζεται αυτό. Γιατί, γιατί χρειαζόμαστε ενεργούς πολίτες και αποτελεσματικά κράτη. Η ενεργοί πολίτες είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί συμμετοχή του δημόσιου τομέα. Εντάξει, μπορεί κανείς να πει ας αφήσουμε τους εμπειρογνώμονες, το κράτος αρκεί να μας στηρίξει λιγάκι. Όχι κράτος, το δημόσιο τομέα, πρέπει να δεσμεύεται. Οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλοι χρειάζονται κάποια νομιμότητα για να κάνουν τη δουλειά αυτή. Γιατί στο κάτω-κάτω είναι προγράμματα ανάπτυξης για τους ανθρώπους. Έπειτα, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των ανθρώπων, γιατί όταν οι άνθρωποι είναι συνειδητοποιημένοι και συμμετέχουν, αυτοί θα κάνουν τη διαφορά με τον τρόπο που ψωνίζουν, με τον τρόπο που ζουν, με τον τρόπο που καταναλώνουν. Πολύ σημαντικό αυτό για να υπάρξει κάποια συστημική αλλαγή. Και αυτά δεν είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι δυνατόν να το πετύχουμε έτσι το στόχο μας. Γι' αυτό και η αναπτυξιακή παιδεία είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθάει τον κόσμο να συνειδητοποιηθεί, να συμμετέχει και είναι μια διαδικασία εκμάθησης αξιών. Κάτι το οποίο είναι βιώσιμο, κρατάει και οδηγεί στην αλλαγή, γιατί ακριβώς αντέχει στον χρόνο. Τώρα συμμετοχή της κοινωνία των πολιτών γιατί, γιατί οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι προκλήσεις μόνο του Νότου, ούτε είναι προκλήσεις μόνο του υποανάπτυξη κόσμου. Όχι, είναι προκλήσεις που έχουν να κάνουν με όλους μας. Οι κλιματικές αλλαγές για παράδειγμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από μερικού μόνο. Απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας. Οι ανισότητες έπειτα και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τοπικά. Και αυτέ για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται τη συμμετοχή όλων. Χρειάζονται μια άλλη γεωπολιτική δομή. Είμαστε στα πλαίσια της ομάδας των 8, ήμασταν μάλλον, τώρα έχουμε φτάσει στους 20-20 συν. Πρέπει λοιπόν να αντιλαμβανόμαστε ότι οι προκλήσεις αυτές είναι παγκόσμιες και άρα χρειάζονται ε, λύσεις στις οποίες να συμμετέχουν όλοι και ο Βορράς και ο Νότος. Όχι μόνο ο Βορράς, μόνο ο Νότος. Νομίζω λοιπόν ότι η αναπτυξιακή παιδεία, και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια, να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική γιατί ακριβώς συνδέει αυτόν που προσφέρει και αυτόν που λαμβάνει. Κάνει αυτή τη σύνδεση. Είναι ένα αδιώνυμο κατά κάποιο τρόπο βοηθάει στο να νιώσουμε όλη την ευθύνη μας και να την μοιραστούμε με αυτούς που χρειάζονται τις λύσεις. Την τελευταία διαφάνεια δεν θα σας την εξηγήσω. Βασικά πρόκειται για τρεις περιπτώσεις, όχι για τόσο νέες. Η αναπτυξιακή παιδεία πρέπει να έχει να προσφέρει κάτι σε όλους τους τομείς. Ανθρώπινα δικαιώματα, υπευθυνότητα, να παίρνει κανείς το μέλλον του στα χέρια του. Η αναπτυξιακή παιδεία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Χωρίς να κάνει διάκριση βορράς-νότος. Πρέπει επίσης να γίνεται μια αξιολόγηση στην αναπτυξιακή παιδεία επικριτική για να δούμε πού είναι οι αδυναμίες και ποια είναι τα δυνατά στη μία. Για να είμαστε σίγουροι ότι η αναπτυξιακή παιδεία προσφέρει. Και θα ολοκληρώσω από τον Τάκαν Ρίν, από το βιβλίο του, που αναφέρει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον 21ο αιώνα και τα βάζει πολύ ομαλέ, ότι ο αιώνας αυτός είναι ένας αιώνα κατά τον οποίο η ανθρωπότητα ή που θα βουλιάξει ή που θα μάθει να κολυμπάει Όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Πρέπει να δούμε όμως ποιος τελικά είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται μαθήματα κολύμπησης και ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει να μάθει κολύμβη στην ανθρωπότητα. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε την σύντομη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο γι' αυτό, αλλά... Η κυρία Σκάλλον. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Με... Μας έδωσαν εικόνα των διαφόρων διαστάσεων του θέματος. Μιλήσατε και για την ατομική εκπαίδευση, τις υπνέπειες που έχει η εκπαίδευση για το άτομο. Είναι σημαντικό να δούμε τις δύο διαστάσεις της εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες που αποκτά το άτομο για να βιώσει στον 21ο αιώνα, αλλά και ο αντίκτυπο τη παιδεία στην κοινωνία, ευρύτερα στην αναπτυξιακή εκπαίδευση. Και αυτή τη διάσταση πρέπει να αναγνωρίσουμε. Είχα μια ερώτηση για την πρώτη παρουσίαση που δυσχεραίνεται λόγω των πολλών ε, διαστάσεων του θέματος. Μπορούμε να μετρήσουμε κατά πόσον έχουμε πετύχει Υπάρχει τρόπος να πούμε αυτό δούλεψε, αυτό δεν δούλεψε. Αυτό που κάνετε στη Φιλανδία για παράδειγμα. Μπορεί να μετρήσουμε τι πετύχαμε για την αλλαγή παλαιών ε, θέσεων για την αναπτυξιακή εκπαίδευση. Έχετε κάνει κάποια έρευνα, μπορείτε. Διότι προφανώ είναι χρήσιμο να μάθει κανεί τι διδαχθήκαμε και τι γίνεται καλύτερα και τι όχι. Κάποιος μίλησε, ανέφερε ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια κοινωνία των πολιτών, αλλά ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. Τα συνδικάτα των εργαζομένων, για παράδειγμα, έχουν ε, μια σειρά δικτύων. Υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση δικτύωσης. Αυτό το να μιλάμε τώρα για Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών είναι και λίγο παρακινδυνευμένο γιατί συχνά η κοινωνία των πολιτών, η ΜΚΟ, δουλεύουν ε, με βάση την εθνική αντίληψη που τους περνάει από τα μέσα, από την κυβέρνηση. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. Πώς θα πετύχουμε την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών. Προφανώς όταν υπάρχουν παγκόσμιες αρμοδιότητες, υπάρχει η εικόνα της ποικιλομορφία. Ναι, αλλά μέχρι... το ερώτημά μου είναι πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Ευχαριστώ κύριε Λόβιν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους ομιλητές. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που μας περιγράψετε. Μια ερώτηση που έχω για την αύξηση αυτή της παγκόσμια έννοια του πολίτη, κάτι πολύ σημαντικό. Η επόμενη, το επόμενο βήμα. Ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν στην σχέση μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Το επόμενο βήμα στην, στα εκπαιδευτικά σας προγράμματα περιλαμβάνεται και τα διεθνή βήματα το επίπεδο που λαμβάνονται οι αποφάσεις σε εκεί δηλαδή που λαμβάνουν οι αποφάσεις διεθνές επίπεδο και τη δυνατότητα που έχουμε να παρέμβουμε για να, δηλαδή προσπαθείτε να προωθήσετε και δραστηριοποίηση σε μια σειρά θεμάτων που δεν είναι πλέον διεθνή αλλά, ε, που δεν είναι εθνικά αλλά διεθνή. Ένα άλλο θέμα που, που αναφέρθηκε από εσά, κύριε Χλαβίτσκοβα, την ανάγκη εκπαίδευσης των ΜΜΕ. Παρεπίπτων, πολύ ενδιαφέρον ωστόσο σχόλιο. Πώς θα το κάνετε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να περάσουμε την επίγνωση αυτή ευρύτερα. Και η τελευταία διαφάνεια του κυρίου, της παρουσίασης του κυρίου Φίλντες μου δημιούργησε μια περιέργεια. Αναφερθήκατε στην ε, έννοια της βοήθειας και ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει αναπτυξιακή βοήθεια. Μπορείτε να μα περιγράψετε κάπως καλύτερα την έννοια αυτή, το, το περιεχόμενο τη τελευταία της τελευταίας Άλλα σχόλια ή ερωτήσει. Όχι. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Χραβίσκοβα. Ναι. Να απαντήσω ειδικά στο ερώτημα για το ρόλο των μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία της ανάπτυξης. Σημαντικό θέμα για μας γιατί προσπαθούσαμε να μην καλύψουμε μόνο την επίσημη εκπαίδευση αλλά και να δούμε την εκπαίδευση της κοινωνίας και του κοινού ευρύτερα και προσπαθούσαμε να περάσουμε στο κοινό με ευκολότερο τρόπο τα θέματα παγκόσμιας εκπαίδευσης ε, με ευκολότερο τρόπο και γι' αυτό για μας, εμάς το Υπουργείο Εξωτερικών δηλαδή τα μέσα είναι πολύ σημαντική παράμετρος για να περνάμε και ειδήσει για τα παγκόσμια ζητήματα αλλά ειδικότερα για την αναπτυξιακή συνεργασία. Πιστεύουμε λοιπόν και χρησιμοποίησαμε την εμπειρία άλλων χωρών της Ευρώπης που είναι πολύ πιο μπροστά από μας τις σκανδιναβικές χώρες για παράδειγμα που έχουν ειδικά προγράμματα όπου χρηματοδοτούν ταξίδια εκπροσώπων των μέσων σε αναπτυσσόμενες χώρες και τους βοηθούν να παράσχουν, να λάβουν πληροφορίες για την κατάσταση της βοήθειας, για την κατάσταση των χωρών αυτών. Επίσης, η γενική διάδοση των ε, πληροφοριών για τη στρατηγική, τις ε, που καλύπτει η στρατηγική αυτή, είναι θέματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη από το ξεκίνημα. Ευχαριστώ. Κύριε Φίτλερ. για το θέμα της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών. Δύσκολο θέμα βέβαια. Ο λόγος ωστόσο που το ανέφερα και που θεωρώ ότι είναι σημαντικός είναι γιατί αμφισβητεί ενιολογικά καταρχάς αυτή τη ε, διαχωριστική γραμμή μεταξύ του εμείς και του αυτή. Είναι μια ιδέα, όχι συγκεκριμένο βήμα στη φάση αυτή. Αλλά για να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ε, βήματα. Η αποτελεσματικότητα των, ε, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η αποτελεσματικότητα αυτών των οργανώσεων γίνεται πολύ μεγαλύτερη όταν μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι ΜΚΟ αυτή τη στιγμή. Τώρα, για την αύξηση της επίγνωσης των πολιτών και τις σχετικές δράσεις. Οι εκπαιδευτές στην ανάπτυξη πάντα τονίζουν ότι το πέρασμα από την επίγνωση στη δράση είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό για τον, τον διδασκόμενο το τι είδους ε, δράση θα λάβουν. Το να τους δίνουμε λοιπόν μία επιλογή δραστηριοτήτων, εκστρατιών κλπ. Είναι σημαντικό για να μπορούν να το διερευνήσουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι και οι διδάσκοντες. Νομίζω για τη βοήθεια. Ε, είναι πολύ σημαντικό να μην ε, αποφύγουμε μια στεναρή συζήτηση για το θέμα της βοήθειας. Γιατί αν δώσουμε την εικόνα ότι δεν μπαίνουμε στη συζήτηση αυτή, χάσαμε το παιχνίδι από την αρχή. Πολλοί εκπαιδευτές στην ανάπτυξη υποστηρίζουν σημαντικά την ένα αποτελεσματικό σύστημα βοήθειας. Αναγνωρίζουν ωστόσο ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για το πώς αναμορφώνουμε τα προγράμματά μας και την αντιμετώπιση τους. Αν δεν τα αντιμετωπίζουμε, τα μεγαλώνουμε. Γι' αυτό ε, τόνισα την ανα... Ε, έχω μια πολύ κριτική στάση στη βοήθεια, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κύριε Ανδρεώτη, ένα μικρό σχόλιο για την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών και τα μέτρα, πολύ σημαντικό, για το Κοινοβούλιο. Δεν θα απαντήσω στο ερώτημα αυτό, θα σας παραθέσω έναν Έλληνα πανεπιστημιακό που μόλις συνάντησα σε μια διάσκεψη για την ευρωπαϊκή ταυτότητα την περασμένη εβδομάδα που, με τον οποίο συζητούσα την κρίση στην Ελλάδα και το τι γίνεται με τους φοιτητέ του που γυρίζουν στα νησιά για να δουλέψουν τα χωράφια και να προστατεύσουν τα νησιά τους διότι θεωρούν ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές πάνε να εξαγοράσουν τα νησιά. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση για το ποιοι είναι υπέρ των νεοφιλελεύθερων, τόσο των εικαζομένων ως νεοφιλελεύθερων πολιτικών και αυτών που είναι αντίθετοι με αυτές τις πολιτικές και υποστηρίζουν την επιστροφή στο κράτος πρόνοιας. Ή τόσο είναι ιδεώδες κράτος πρόνοιας. Ήταν ο πρώτος που ρώτησε σε μια ευρωπαϊκή διάσκεψη ποιος το πληρώνει Ποιος την πληρώνει την πρόνοια. Υπάρχει ένα γλυπτό ενός ε, δανού γλύπτη, μιας πολύ παχιάς γυναίκας, ε, στην πλάτη, που, που, στηρίζεται στην πλάτη ενός αδύναμου Αφρικανού και του λέει θα κάνω ό,τι μπορώ να σε βοηθήσω πλην του να κατέβα από την πλάτη σου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και καθώς η κρίση εξελίσσεται μπορεί να μην έχουμε επιλογή όπως είπε και ο Ματίας πρέπει να μάθουμε να κολυμπούμε όλοι μαζί. Το θέμα λοιπόν μιας παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών δεν είναι μόνο η δημιουργία της, αλλά και η εμπλοκή της στο πολύ σύνθετο πλαίσιο στο οποίο δουλεύουμε. Τώρα, το θέμα της μέτρησης όντως είναι πολύ σημαντικό για οικονομικά ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ένα μοντέλο. Αξιοποιούμε και αποτιμούμε μόνο ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε. Τώρα πρέπει να μπορούμε να μετρούμε, να αλλάξουμε μορφή, να αλλάξουμε προσέγγιση και να μετράμε αυτό που, αποτι... που θεωρούμε σημαντικό. Ας πούμε, στην κινητικότητα πρέπει να αρχίσουμε να αποτινούμε και οικονομικά και κοινωνικά την κινητικότητα. Το να στέλνεις κάποιον σε διάφορες χώρες, το να δημιουργήσεις αυτή την παγκόσμιότητα, την παγκόσμια ηθαγένεια, ε, πόσο κοστίζει, πόσο προσφέρει. Πιστεύω ότι μεθοδολογικά οι δομές αυτές είναι σωστές, αλλά θεωρητικά ε, δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, για την τόσο σημαντική συζήτηση. Και ε, δίδω τον λόγο εις ε, τον ε, κύριο Νόισερ τον, θέλω να σας α, συγχαρώ όλους ε, για το σεβασμό του χρόνου σας και ε, πριν ξεκινήσει η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα ήθελα να σας πω ότι όπως και ο κύριος Πίμπαλξ ήμουνα και εγώ ο ε, καθηγητής και διευθυντής σε σχολείο και ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπω τους νέους οι οποίοι προχωρούσαν προς ένα καλύτερο κόσμο εδώ θα συζητήσουμε την στρατηγική για μια ευρωπαϊκή αναπτυξιακή παιδεία και ε, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των κρατών μελών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τέλος ε, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους μηχανισμούς για να προωθήσουμε πιο αποτελεσματικές επεμβάσεις. Ε, επίσης θα αναλύσουμε τα υπέρ και τα κατά της παρούση στρατηγική για να καταλάβουμε καλύτερα πόσο η αναπτυξιακή παιδεία μπορεί να συμβάλλει σε ένα νέο ε, αναπτυξιακό παράδειγμα, δηλαδή ε, μία πολιτική συνεκτικότητα για την ανάπτυξη, για την αποτελεσματικότητά της και για τα ανθρώπινα δικαιώματα που βασίζονται στην ανάπτυξη. Ε, πέραν αυτού θέλουμε να προωθήσουμε ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως της πολιτικής και της στρατηγικής της και των σχετικών πολιτικών των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων διότι σε πολλά κράτη-μέλη αυτή η συνεργασία δεν υπάρχει ακόμη και θα δώσω καταρχήν τον λόγο τον Κρίστοφ Στανόφσκι τον οποίον παρακαλώ αν είναι δυνατόν να καλύψει το θέμα του σε 10 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνει γίνεται. Η ε, παιδεία στην Πολωνία θεωρείται πολύ σημαντική και καλύπτει τουλάχιστον τον 1 πέμπτο της ε, χώρας ε, διότι πριν από 10 χρόνια ήμασταν οι πρωταθλητές αλλά πριν 3 χρόνια ήμασταν πρωταθλητές ε, πριν από 30 χρόνια ήμασταν πρωταθλητές ε, για να ε, απορρίπτουμε την κυβέρνηση και να αρνούμαστε και έτσι δημιουργήθηκε η Σολιντανόσκ. Και 10 χρόνια μετά η κυβέρνηση, το κράτος αλλά και εμείς καταλάβαμε ότι δεν φτάνει να αντιστακόμαστε έπρεπε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας προς ε, τις ε, κοινωνίες των πολιτών για την τοπική αυτοδιοίκηση και μετά μερικά χρόνια ε, μπορέσαμε να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σήμερα έχουμε την Προεδρία και είμαστε μία από τις χώρες δωρητές για την συνολική αναπτυξιακή συνεργασία και την παιδεία και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά συγχρόνως ε, και ε, ε, στον παγκόσμιο χώρο. Κατά κάποιο τρόπο έτσι περιγράφεται η συνολική παιδεία. Πρέπει δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι δεν φτάνει να αντιστεκόμαστε και να διαμαρτυρόμαστε αλλά πρέπει η συνολική κοινότητα να προχωρήσει περαιτέρω πέρα των των εθνικών συνόρων και αυτό που μας απασχολεί ε, όταν συζητάμε για την παιδεία και για την Πολωνία είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο τελικός στόχος είναι να συμμετέχουν στην προσπάθεια και οι πολίτες να είναι καλά κατηρτισμένοι, καλά προετοιμασμένοι και να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά και να εμπλακούν άμεσα στην αναπτυξιακή συνεργασία. Βεβαίως πρέπει να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις, θα πρέπει να υπάρχει μία καλύτερη συνολική παιδεία και αυτό είναι κάτι το οποίο επετεύχθη τα τελευταία χρόνια διότι όπως όλοι οι τομείς της παιδείας στην Πολωνία συνέβαλαν στο θέμα αυτό οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και εγώ ήμουν ένας από τους αρχηγούς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Πολωνία και δίδασκα ότι η πολιτική παιδεία πρέπει να συμβάλλει στην συνολική η εκπαίδευση και ε, η χώρα μας κατάφερε να ε, ε, αναβαθμίσει τη συνολική παιδεία και αυτό επετεύχθη στη χώρα μας σε κάθε επίπεδο της, του εκπαιδευτικού χώρου και τέλος απετέλεσε έναν σημαντικό τομέα ή στην κατάρτιση των διδασκόντων και αυτό που είναι σημαντικό σε αυτό το τομέα είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να μην αποκλίνονται να μην αποκλείονται από τα αποτελέσματα δηλαδή ένα σημαντικό μέρος του ότι ε, ε, διεξάγεται στην αίθουσα της διδασκαλίας επηρεάζεται από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θεωρήσαμε λοιπόν αυτό πολύ σημαντικό δηλαδή ότι οι κυβερνητικές οργανώσεις έπρεπε να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει για μας. Δηλαδή πολλές χώρες οι οποίες εξέτασαν το τι κάναμε και μας στήριξαν πολύ και στην κίνηση αυτή στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος μπορέσαμε να καταρτήσουμε με τα πτυχιακά προγράμματα για τους διδάσκοντες και για πρώτη φορά η Πολωνία έχει καταρτήσει νομοθεσία ε, όπου η ε, συνολική ε, συνεργασία στον τομέα της παιδείας κατοχυρώνεται. Θεωρούμε ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο, αλλά υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων και αυτή η διαδικασία του διαλόγου μεταξύ των συνεργατών είναι πολύ σημαντική για να αναπτύξουμε τη δική μας στρατηγική διότι το Υπουργείο του ε, το Υπουργείο ε, συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών, ε, το Υπουργείο Επιστημών και είναι σημαντικό ότι τα προγράμματα που καταρτίζονται απευθύνονται ή στους διδάσκοντες, στα σχολεία, στους μαθητές, ε, στα μέσα ενημέρωσης και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τα μέσα ενημέρωσης είναι σημαντικά για να επικοινωνούμε και προς ε, την κοινωνία, προς το ευρύτερο κοινό αλλά και προς τους διδάσκοντες και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μία σωστή κάλυψη του ε, τι γίνεται στον τομέα της παιδείας. Είναι μια σημαντική ε, στιγμή για την ανάπτυξη της συνολικής παιδείας εις ε, την Πολωνία διότι υπεγράφει ε, μία συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας ε, της Ενώσεως των Πολωνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ένα μνημόνιο το οποίο ε, περιλαμβάνει και τους ορισμούς αλλά και τα σημεία συμφωνίας σχετικά με το πώς θα διεξαχθεί αυτή η συνεργασία. Όταν σκεφτόμαστε την συνολική παιδεία πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Κίνας, της Ρωσίας, της Τουρκίας, της Βραζιλίας. Υπάρχει κάποια διαφορά. Εγώ διαπιστώνω μία ουσιαστικά και αυτό είναι η συνολική σφαιρική παιδεία. Δηλαδή το να κατανοήσουμε ότι η Ρωσία πριν από λίγες μέρες μόνο κατήρτισε μία αναπτυξιακή οργάνωση και γνωρίζοντας τη Ρωσία δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσουν προς μία σφαιρική παιδεία. Κατά κάποιον τρόπο αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε ήδη αναπτύξει στην Ευρώπη. Είναι κάτι μοναδικό το οποίο πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει μόνο να επενδύουμε στο νότο να βοηθήσουμε την οικονομική προσπάθεια και την ανάπτυξή τους αλλά ότι πρέπει συγχρόνως να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να εξουσιοδοτήσουν τις τοπικές κοινωνίες για να μπορεί να υπάρχει αυτοδιάθεση του λαού και ε, να ε, μπορέσει ε, ο λαός να κατανοήσει το τι κάνουμε όχι μόνο σαν αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά πρώτα και πρωταρχικά στο επίπεδο των πολιτών και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σφαιρικής συνολικής παιδείας και έτσι υπάρχει ενημέρωση για να στηριχθεί η ανάπτυξη όχι μόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια και, ε, αλλά στην ε, δημιουργία μιας, ε, ενός θεσμού Ευρωπαίων πολιτών διότι αυτό το είδα προημερών με την, με την Επίτροπο Γεωργίευα και είδαμε ότι αυτό που έλειπε στην εκδήλωση που οργάνωσε ήταν μια ευρωπαϊκή σημαία. Μείναμε λοιπόν λοιπόν στην εκδήλωση αυτή ε, μια ολόκληρη μέρα και είδαμε μόνο κάποια στιγμή μια ευρωπαϊκή σημαία πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν προβαλόμεθα επαρκώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό κατακρίνεται ότι δεν βοηθά επαρκώς και συγχρόνως δεν περνάμε το μήνυμα προς τους ενδιαφερόμενους για το τι έχουμε κάνει και επίσης το μήνυμα αυτό δεν μεταδίδεται καν στους πολίτες μας ότι δηλαδή εμείς μπορούμε κάτι να κάνουμε το οποίο να είναι πραγματικά σημαντικό. Συνήθως το, η επόμενη ερώτηση είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα και το επόμενο βήμα καταρχήν πρέπει να είναι το θέμα του εάν μπορούμε μεταξύ κρατών μελών να συζητάμε περισσότερο για θέματα παιδείας. Εάν η συζήτηση για την συνολική παιδεία, την πολιτική παιδεία μπορεί να βοηθήσει στην κατάρτιση κοινών προδιαγραφών και να μην έχουμε μόνο προδιαγραφές για τα μαθηματικά και ίσως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Και τέλος, το τελευταίο μου θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να κινηθούμε από την συνολική παιδεία προς την δράση. Ένας τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο ε, είναι κάτι που ήδη ανέφερα προ λίγων λεπτών. Δηλαδή καινοτόμα οικονομικά μέσα τα οποία οι υπάρχουν ή ε, την Πολωνία, στην Τσεχία και σε άλλες χώρες, δηλαδή τον νόμο του 1%, το δικαίωμα 1% της φορολογίας ε, να ε, χρησιμοποιηθεί για την παιδεία και αυτό έχει τη στήριξη του κοινού διότι οι φόροι αυτοί θα μπορούν να διοχετευτούν προς ανθρώπους που χρειάζονται χρειάζονται βοήθεια στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Πολωνία που κινούνται εν ονόματι των πολιτών και προσαρμόζονται στις ανάγκες των πολιτών και όχι στις επιταγές των πολιτικών και μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά να βοηθήσουν ή στο να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Στενόφσκι. Επαναλαμβάνω ότι για μένα το βασικό θέμα για την παγκόσμια εκπαίδευση είναι ότι πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίζουμε αυτό όλοι οι Ευρωβουλευτές. Ο Helmut Χαρτμάγερ έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Χαρτμάγερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να έρθω σε αυτήν την τόσο δικαικριμένη και σημαντική νομίζω συνεδρίαση. Με ιδιαίτερη χαρά μιλάω μετά από τον ε, συνάδελφο και φίλο, μπορώ να πω, Στανόφσκι και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Με ιδιαίτερη χαρά. Επίσης συμμετέχω και εγώ ως δάσκαλος στην αίθουσα αυτή, γιατί και εγώ ήμουν δάσκαλος για καιρό. Και νομίζω ότι όντως λίγο πολύ αισθάνομαι σαν μέσα σε μια τάξη εδώ. Θα σας μεταφέρω λίγο τους προβληματισμούς μου για μια ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης της παγκόσμιας εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι χρειάζεται πραγματικά μια τέτοια πολιτική για την αναπτυξιακή παιδεία στην Ευρώπη και πρέπει να έχουμε μια καλή βάση. Και νομίζω ότι υπάρχει. Έγινε μια μελέτη πέρυσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αναπτυξιακή Παιδεία και τη συνειδητοποίηση και την Ανάπτυξη και η μελέτη αυτή όσον αφορά τις διάφορες έννοιες, καταλήγει σε δύο συστάσεις. Πρώτον, να χρησιμοποιούμε τον όρο παγκόσμια μάθηση, global learning, γιατί όντως πρέπει να είναι μια άσκηση μάθησης. Και υπογραμμίζει επίσης και τη σημασία που έχει η δράση παρέμβασης, advocacy work, campaigning, να αποτελεί κάτι σαν εκστρατεία, γιατί πρέπει να καταλήγουμε σε μια δράση. Και αυτό αναφέρθηκε και νωρίτερα με κάποια διαφάνεια. Αυτό που μπορούμε να μάθουμε λοιπόν από τον κύριο Φίλερ είναι ότι πραγματικά χρειάζεται προβληματισμός και δράση, ένας καλός συνδυασμός των δύο αυτών ενιών. Ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια με μια μεγάλη διάσκεψη που οργανώθηκε στην Ολλανδία στο Μάστριχτ από το Συμβούλιο της Ευρώπης και στη διάσκεψη αυτή ε, καταλήξαμε σε μία δήλωση στο τέλος. Και η δήλωση αυτή λέει ότι η παγκόσμια εκπαίδευση η εκπαίδευση για την ανάπτυξη δηλαδή είναι κάτι το οποίο ανοίγει τα μάτια και το μυαλό του κόσμου σε πραγματικότητες του κόσμου και τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ε, την ανάγκη για περισσότερη δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό περιεχόμενο αυτό για τη στρατηγική που πρέπει να αναπτύξουμε. Είναι μια στρατηγική που πρέπει να βασίζεται στο περιεχόμενο στο περιεχόμενό της βάσει μιας πολυατομικής προσέγγισης. Δηλαδή πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την ε, εκπαίδευση για την ανάπτυξη και την διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αηφόρο ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και να συμμετέχουν σε αυτό διάφοροι παράγοντες. Και χάρηκα από ο κύριος Πίπελς νωρίτερα είπε πως μια τέτοια ευρωπαϊκή στρατηγική συμπληρώνει τις ε, δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλοί εθνικοί παράγοντες, οι διάφορες κυβερνήσεις, τα Υπουργεία, η εκπαιδευτική κτλ. στι διάφορες χώρες. Και είναι πολύ σημαντική και η δουλειά που γίνεται από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις βέβαια. Για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τώρα την εμπειρία που διαθέτουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, φτιάξαμε ένα δίκτυο. Το ακούσαμε και νωρίτερα σήμερα το πρωί. Το δίκτυο αυτό ονομάζεται GIN. Είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Παγκόσμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν εθνικά υπουργεία, οργανώσεις και διάφοροι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την στήριξη και για την εκπόνηση πολιτικής σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παγκόσμια εκπαίδευση και εκμάθηση. Πρόκειται για 31 μέλη, πρόκειται δηλαδή για, μια, για ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν από 20 χώρες 31 ε, διαφορετικές οργανώσεις. Με σύνολο 100 εκατομμύρια ευρώ. Η βάση για το δίκτυό μας αυτό είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε με μια πρόσθετη αξία από το δίκτυό μας. Και αυτό είναι ότι διευκολύνουμε, ε, για παράδειγμα, να μπορούμε να έχουμε μια συγκριτική εκμάθηση. Έπειτα να γίνεται μετάδοση των ε, στρατηγικών που έχουμε σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη, να τις μεταφέρουμε και αλλού δηλαδή. Έπειτα επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα, στην αξιολόγηση και στη βελτίωση. Επίσης στην μετάδοση πληροφοριών, να τις μοιραζόμαστε δηλαδή με τους άλλους ό,τι πληροφορίες ε, έχουμε για σωστές πολιτικές. Γίνεται αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων και συμμετέχουμε και σε επίπεδο ε, εκμάθησης και ε, εκπαίδευσης που βγαίνει κάπως από τα επίσημα σχολικά προγράμματα. Στην ε, χώρα μου, μια από τις συστάσεις που έγινε με την αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων ήταν να φτιάξετε μια εθνική στρατηγική. Και το κάναμε με το Υπουργείο Παιδείας αναπτύξαμε μία στρατηγική για την παγκόσμια εκπαίδευση και το συμπεριλάβαμε στο σχολικό πρόγραμμα. Και ενισχύσαμε λοιπόν την αναπτυξιακή παιδεία και φροντίσαμε να υπάρξει παρετέρω έρευνα έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη των διαφόρων ενιών στον τομέα αυτό και τώρα ετοιμάζουμε μία στρατηγική και για ε, την ε, μη επίσημη εκπαίδευση, δηλαδή την εκπαίδευση που προσφέρεται εκτός σχολικών προγραμμάτων στα παιδιά και στους νέους. Πολύ σύντομα τώρα θα θίξω λίγο τις εμπειρίες που έχουμε σε εθνικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν πολλές και θα μπορούσαν να υπάρχουν και πολύ περισσότερες για να αναφέρουμε εδώ. Η Τσεχία είναι ένα παράδειγμα από ό,τι έμαθα και άκουσα, η Σλοβακία επίσης. Έχουμε στρατηγικές τέτοιες επίσης και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα στη Φιλανδία και στην Ιρλανδία. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα που αναφέρω. Και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση προκειμένου να αναπτύξουμε και μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Πώς τώρα όμω να αναπτύξουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή στρατηγική. Θα σας κάνω κάποιες συστάσει που βασίζονται στη δικιά μας εμπειρία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα διαφερόμενα μέρη. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα που ακριβώς να δείχνει ποιοι συμμετέχουν και ποιος κάνει τι, διαφάνεια δηλαδή. Τρίτον, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Πρέπει να, δίνουμε, να προσφέρουμε στον εαυτό μας το χρόνο που χρειάζεται ώστε να αναπτύξουμε ε, την ε, σωστή στρατηγική με αποφασίζοντας ποιος θα αναλάβει τον ηγετικό ρόλο. Έπειτα πρέπει να διασαφηνίσουμε ε, τις έννοιες και να βρούμε και να χρησιμοποιήσουμε συμμαχίες για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και τέλος, πρέπει την ανάπτυξη μιας τέτοια στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής δηλαδή, ε, να το δούμε σε κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζεται. Ισαΐ. Είναι ένα καλό μήνυμα αυτό πιστεύω, το να το δούμε έτσι σαν ε, μια στρατηγική εκμάθηση, χρησιμοποιώντας βέβαια τις υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές και εμπειρίες. Να χρησιμοποιήσουμε την αξιολόγηση, όπως σας είπα πριν, μεταξύ ομοτήμων, να χρησιμοποιήσουμε προγράμματα που μας έρχονται από τα νέα κράτη-μέλη και που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα και τέλος να λάβουμε υπόψη μας τις συστάσεις της μελέτης DEAR που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα έπρεπε να περιλαμβάνεται τώρα μέσα σε μια τέτοια ευρωπαϊκή στρατηγική. Πρώτα απ' όλα να έχουμε ξεκάθαρους ε, στόχους στρατηγικής να καθορίζονται σαφώς οι προτερότητες επίσης, γιατί δεν μπορεί να καλύψουμε όλα τα θέματα μια και έξω. Πρέπει να υπάρχει μια πρόσθετη αξία για τις πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη. Μίλησα πριν για τη συμπληρωματικότητα μιας τέτοιας στρατηγικής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει επίσης μια ευρωπαϊκή στρατηγική να οδηγεί στην ενίσχυση του συντονισμού με τα κράτη-μέλη. Να υπάρχει διάλογος δηλαδή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Θα έπρεπε επίσης να υπάρχουν ε, συναντήσεις με όλα τα κράτη-μέλη και με τους πιο βασικούς ε, παράγοντες και τέρους συχνά. Να ενισχύσουμε επίσης και ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις αλλά και παγκόσμιες έτσι ώστε να αποτελεί μια πραγματικά διεθνή άσκηση η στρατηγική αυτή. Και τέλος, να ενισχύσουμε στα κράτη-μέλη, δύο στα νέα κράτη-μέλη, αυτό που ονομάζουμε capacity building, δηλαδή ε, οικοδόμηση ικανοτήτων. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα εδώ και περιμένω να συμμετάσχω και στις μελλοντικέ συζητήσεις για το θέμα. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαρτμαγερ. για τον σαφή λόγο σας. Υπογραμμίζω αυτό που είπατε. Η μάθηση σημαίνει και σκέψη και δράση. Ο κ. Ντένις Χούμπερ το έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα απομακρυνθώ από τις σημειώσεις ε, που έχω ετοιμάσει και που είναι στη διάθεσή σας προσπαθώντας να σκεφτώ και να δουλέψω αυτά που ήδη αναφέρθηκαν. Δύο λόγια καταρχάς για το κέντρο Βορανότου. Μπορεί να μην το ξέρετε όλοι. Το κέντρο μας δημιουργήθηκε πριν από 21 έτη όταν έπεφτε το τείχος του Βερολίνου. Ο στόχος τότε του κέντρου αυτού ήταν να προωθήσει την παγκόσμια ελεξάρτηση και αλληλεγγύη μεταξύ των πληθυσμών της Ευρώπης για να εξασφαλίσει ότι ο Νότος δεν θα ξεχαστεί σε μια στιγμή που όλοι κοίταζαν ανατολικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολύ πρόσφατα, το Μάιο του 11, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, υιοθετήθηκε ένα νέο καταστατικό ψήφισμα για το κέντρο του νότου από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπεβεβαίωσε τη σημασία του στόχου αυτού. Ακούσαμε βέβαια να λένε πολλοί ότι γίναν πολλά, πολλά μένουν να γίνουν, αλλά υπάρχει και ένα νέο, ένας νέος στόχος που μπορούμε να εξετάσουμε, να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία έξω από την Ευρώπη, πέραν των ορίων της Ευρώπης, ιδίως στις γειτονικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Προφανώς το ψήφισμα αυτό συνδέεται, όπως καταλαβαίνετε, και με, το λεγόμενο, με τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Το κέντρο Βορανότου είναι ένας θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά έχει και ισχυρή κοινοτική, ενωσιακή συμμετοχή, όπου και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και προ πρόσφατα και η Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Βορανότου. Είναι ένα σπάνιο σχετικά παράδειγμα λοιπόν όχι μόνο ουσιαστικής συνεργασίας αλλά και θεσμική συνεργασίας μεταξύ δύο δομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ακόμα να κάνουν βήματα για να τα βρουν απόλυτα. Τώρα, να σας αναφέρω κάποιες ιδέες που έχω θα αναφερθώ σε μία φράση του Αβραάμ Λίνκολν που έλεγε πριν αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού είμαστε. Πρώτα λοιπόν, από πού προερχόμαστε. Πολλά αναφέρθηκαν ήδη και θα είμαι σύντομος. Ερχόμαστε μετά από μία δεκαετία εντατικής δουλειάς, αύξηση της επίγνωσης και προώθησης της νέας εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω των ε, δομών της συνεργασίας. Δύο παράμετρους θα αναφέρω. Η διάσκεψη του Μάστριχ το 2002, το είπε και ο γείτονά μου, υιοθέτησε ένα πρόγραμμα δράσης μέχρι το 2015 και το Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση, μια προσπάθεια στην οποία μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και που οδηγεί, στοχεύει στον οδηγεί σε μια συνένεση για το τι σημαίνει αναπτυξιακή εκπαίδευση και τι στόχο έχει. Το ενδιαφέρον που βλέπουμε όταν ρωτάμε από πού ερχόμαστε είναι ότι ερχόμαστε από ένα πολύ σύνθετο πλαίσιο με πάρα πολλούς ενεργούς διαφορετικούς φορείς. Μία λοιπόν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, κοινή πρόκληση και που πιστεύω ότι είχαμε καλά αποτελέσματα ήταν η συνεργασία. Κάτι που δεν ήταν αυτονόητο πριν από 10 χρόνια. Πολλοί θεσμοί, η Ένωση, το Συμβούλιο, κάνουν τις δικές τους δουλειές, δεν συνεργάζονται πάντα και κράτη-μέλη ωστόσο, υπογράμμισε ο γείτονά μου τη σπουδαιότητα της συμπληρωματικότητα μεταξύ του τι επιτυγχάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών, το δίκτυο είναι πολύ σημαντικό στη διαδικασία αυτή, αλλά βεβαίως προφανώς ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης καθοριστικός. Ο εξαριστερών ε, συγκαθήμενός μου παίζει καθοριστικό ρόλο σε μία από αυτές τις πλατφόρμες. Θα σας μιλήσει γι' αυτό φαντάζομαι. Μια λοιπόν βασική πρόκληση ήταν η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια και νομίζω με τα τελευταία 10 χρόνια κάναμε καλή δουλειά σχετικά. Πού βρισκόμαστε τώρα, σήμερα. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου όχι μόνο πετύχαμε καλύτερη συνεργασία, αλλά και θεσμοθετημένη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που έχει πολιτική και οικονομική υποστήριξη από την Επιτροπή, κάτι πολύ σημαντικό και αυτό θα ήθελα πραγματικά να υπογραμμίσω και να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την υποστήριξή της. Υιοθετήθηκαν πρόσφατα εθνικές στρατηγικές σε πολλά κράτη-μέλη, ιδίως νέα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά και την Πορτογαλία, τη χώρα από όπου προέρχομαι, όχι εγώ δηλαδή, όπου, προέρχεται, όπου είναι εγκατεστημένο το κέντρο βορανότου, ξέχασα να σου το πω. Στοχευμένες προσπάθειες κάνουμε στα νέα κράτη-μέλη της Ένωσης, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και Μεσόγειο, την Κύπρο, τη Μάλτα. Κάναμε ειδική προσπάθεια μέσω μιας κοινή ε, συμφωνία, διαχειριστικής συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ Επιτροπής και Κέντρου Βορανότου. Ο στόχος της συμφωνίας αυτής για την περίοδο 9-11 ήταν, βρισκόμαστε λοιπόν στο τελευταίο έτος εφαρμογής αυτής της κοινή συμφωνίας. Επίσης, η μελέτη ΔΕΑ που δείχνει πολύ σημαντική γιατί δείχνει τι πετύχαμε, αλλά δίνει και παρουσιάζει και κάποιες συστάσεις για τις προτεραιότητες που θα πρέπει να υιοθετήσουμε στο μέλλον. Πρόσφατα δε εγκρίναμε το πρώτο ευρωπαϊκό νομικό πρότυπο παγκόσμιας εκπαίδευσης μετά από σύσταση του Συμβουλίου των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε πριν λίγους μήνες, το Μάιο του 2011. Για όλα αυτά, και έχω στο τελευταίο λεπτό μου, τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, να χρησιμοποιήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε ό,τι έχουμε ήδη κάνει, που είναι και Δεύτερον, να διευρύνουμε την γεωγραφική μας εμβέλεια. Υπάρχει σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης που τώρα έχει στα σε 47 κράτη-μέλη ε, του Συμβουλίου. Επίσης μπορούμε να δώσουμε έμφαση στις γειτονικές χώρες, κάποιες από τις οποίες όπως το Μαρόκο μετέχουν και στο κέντρο βορανότου. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες να παράσχουμε, να ενσωματώσουμε την παγκόσμια εκπαίδευση στην ε, κανονική εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφέρθηκε από τον, τον Πολωνό Υφυπουργό την ε, σημασία, πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο και τι έκαναν στην Πολωνία, αλλά δυστυχώ η Πολωνία δεν είναι το σύνηθε, είναι η εξαίρεση. Λίγες χώρες έχουν ενσωματώσει αυτή την πολιτική ε, στο εκπαιδευτικό του σύστημα, άρα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο με τα Υπουργεία Παιδείας. Επίσης, Τέταρτη σημασία, συνέχιση του, της σύνδεσης μεταξύ παγκόσμιας εκπαίδευσης και δικαιωμάτων ανθρώπου. Όχι μόνο για να αυξηθεί η επίγνωση για τη σημασία της ανάπτυξης, αλλά γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση, όπου τα ακραία πολιτικά κόμματα έχουν όλο και μεγαλύτερε εκλογικέ επιτυχίες και γι' αυτό θα πρέπει να συνδέσουμε τις προσπάθειές μας με τις προσπάθειες που γίνονται ευρύτερα στην εκπαίδευση για τα δικαιώματα των ανθρώπου. Τελευταία παρατήρηση, να έχουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ευθύνη των πολιτών, διότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε το ότι δεν έχουμε μόνο δικαιώματα αλλά και ευθύνες προς την κοινωνία, προς τον πλανήτη και προς τις νέες γενναίες. Κλείνω. Και θέλω να σας αναφέρω ότι το κέντρο το Μάιο του 12 θα οργανώσει μια πανευρωπαϊκή διάσκεψη στην οποία θα μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να υιοθετήσουμε ένα σχέδιο δράσης για την περίοδο 2011 έως 2015. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χούμπερ και τέλος θα ήθελα να ακούσω τον ε, Λίλι Λαπανάινεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ και πρέπει να σας πω ότι αντιπροσωπεύω πάνω από 16.000 εδώ στην Ευρώπη και έχω ε, θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα. Πρώτον, τις ε, ε, διάφορες τους διάφορους στόχους μας και το μέλλον. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις διότι προ 10 χρόνια το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε σαφώς διατυπώσει πώς θα ήθελε να διαμορφωθεί η αναπτυξιακή παιδεία στο μέλλον και ε, ήταν ε, ένα πολύ ε, καλό θέμα το οποίο ξεκίνησε αλλά το έγγραφο το οποίο καταρτήθηκε και υπεγράφει δεν ήταν δεσμευτικό. Όπως ξέρετε υπάρχει μία συμφωνία η οποία έχει ξεκινήσει το 2005 αλλά από τη δικιά μας άποψη η γνώμη μας είναι ότι ε, χρειάζεται να έχουμε ε, μία πιο σαφή εικόνα και η βασική διαδικασία έγινε κατά την Φιλανδική Προεδρία το 2006. Δεν ε, ε, στηρίχτηκε από τον Επίτροπο Λουί Μισελ και ε, από τους αρχηγών, αρχηγούς κρατών στην Λισαβόνα. Το έγγραφο όμως αυτό περιλαμβάνει διάφορες συστάσεις για διάφορους συμμετέχοντες και βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι ε, ε, εμπλεκόμενοι και γι' αυτό θεωρείται ένα πολύ βασικό έγγραφο στον τομέα αυτό. Δεν ήταν όμως όπως είπα ένα πολιτικά δεσμευτικό έγγραφο Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προβεί σε ε, διάφορες ε, διατυπώσεις και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναφερθεί και πρέπει να αντιληφθούμε γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει όμως να πούμε ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε μία συνολική στρατηγική και πρέπει καταρχήν να έχουμε μία σαφή εικόνα όπως είπαν διάφοροι από τους συναδέλφους Παραδείγματος χάρη, μία διαδικασία δημοσίων ε, σχέσεων οδήγησε στο ότι θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ε, η αναπτυξιακή παιδεία δεν θεωρείται σαν ε, μία κίνηση δημοσίων σχέσεων αλλά προωθεί συνολικά την εκπαίδευση πρέπει όμως πέραν αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μία δικιά της ιδέα και ένα δικό της πρόγραμμα για την παιδεία και θεωρούμε ότι είναι ένα τομέας πολιτικής που είναι πολύ σημαντικός για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μακροπόθεσμα ε, όσον αφορά την οργάνωση των χρηματικών πόρων οι οποίοι θα αφιερωθούν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Τρίτον, ε, Τώρα που διατυπώνεται το νέο πρόγραμμα πλαίσιο, οικονομικό πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει μία μακροπρόθεσμη προοπτική για τις δραστηριότητες της πέραν ε, του ετησίου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπον ώστε αυτή η κοινωνία των ε, πολιτών ε, να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Χρειαζόμαστε συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων ε, και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν οι σωστές ε, πηγές χρηματοδότησης και οι ε, διαδικασίες και δραστηριότητες να έχουν σχέση με την κοινωνία των πολιτών και να παρακολουθούνται από τις αρμόδιες ε, ε, Γενικές Διευθύνσεις Παιδείας και Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα με τους διαφόρους άλλους ε, συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος ε, θα πρέπει να υπάρχει μία ποιοτική αξιολόγηση της παιδείας κατά τρόπον ώστε να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των δράσεων και θα διευκολύνει ε, ε, την πρόθεση της παιδείας. Ποια θα είναι η πρώτη μορφή αυτού του προγράμματος. Έχουμε μία πρώτη ιδέα, διότι πιστεύουμε ότι μία καλή ιδέα θα είναι να υπάρξει μία μία κίνηση ε, η οποία θα αποδείξει τις, ε, τους στόχους και θα μπορέσει να ε, αναφερθεί σε όλες τις δραστηριότητες ε, ξεπερνώντας την μεμονωμένη γραμμή του προϋπολογισμού που αφιερώνεται στο θέμα αυτό. Θα μπορούν ε, οι ενδιαφερόμενοι να ε, επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους στόχους, να υπάρξει συνεκτικότητα, συντονισμός και συνεργίες μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, των κρατών μελών που θα συμπληρώνουν τις προσπάθειες ε, για να υπάρχει μία διαχείριση των γνώσεων και ε, ποιοτική παιδεία καθώς και συνολικές πρωτοβουλίες. Ε, τέλος, ε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ο οποίος να επιτρέπει να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν των δραστηριοτήτων. Θα ήθελα να αναφερθούμε στα βασικά θέματα για να μπορέσουμε μπορέσουμε να α, διατυπώσουμε προτάσεις ε, στις οποίες θα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Ε, θα πρέπει να συντονίζεται η κοινωνία των πολιτών ε, στα θέματα αυτά, να υπάρχει κοινή προσπάθεια για την πρόθεση της παιδείας και καλό θα ήταν να μιλήσουμε και για τη συνολική κοινωνία των πολιτών μια τέτοια στρατηγική η οποία βασίζεται στις προτάσεις της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, συζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αποτελεί μια σημαντική πρόοδο για την πρόωθηση της παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ θα ήθελα να επανέλθω στο γεγονός ότι έχουν προωθηθεί πολύ καλά πολλά ψηφίσματα και θέσεις και αυτό το οποίο ε, λείπει είναι μόνο ένα πολιτικά δεσμευτικό έγγραφο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαπαλάινεν. Πριν δώσω το λόγο στους συμμετέχοντες εδώ, πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Κρίστιαν Σμιτ που είμαι ο νέος διευθυντής ε, για την ε, ε, ανάπτυξη κοινωνίας και ανθρώπων. Έχω να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα για τη στρατηγική και μετά για το περιεχόμενο, μετά από τις διάφορες παρεμβάσεις που ακούσαμε εδώ. Ακούσατε το πρωί τον Επίτροπο Πίμπαλ πρώτα απ' όλα, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η στρατηγική μας, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την μελέτη DR. Έχει πολύ σημασία αυτό και εν ώψη των προτάσεών μας για τις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές, όπου θέλουμε να αυξήσουμε το ποσό για την κοινωνία των ε, πολιτών κατά 20%. Κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε περισσότερα στον τομέα αυτό. Έπειτα όσον αφορά την στρατηγική τώρα και την διαδικασία στήριξης. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Επίτροπος, ε, θα Δημοσιεύσουμε ήδη μια πρόσκληση για προσφορές, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ε, μεγαλύτερο αντίκτυπο και στα πλαίσια αυτά ακριβώς θέλουμε να προσπαθήσουμε να ε, θέσουμε ε, σε εφαρμογή και όλες αυτές τις συστάσεις που έχουμε και από τη μελέτη αλλά και από εσά σήμερα. Ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα μας αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα η σχέση που πρέπει να υπάρχει με ε, το σχολικό πρόγραμμα, με τις σχολικές σπουδές. Να συμπεριλάβουμε δηλαδή την παγκόσμια εκπαίδευση και στο σχολικό πρόγραμμα των κρατών μελών. Δεύτερον, όπως ανέφερε και ο τελευταίος ομιλητής, πρέπει να διευκολύνουμε τη σχέση ανάμεσα σε αυτούς που προσφέρουν και σε αυτούς που παίρνουν. υπάρχει μια καλή διαχείριση της ε, γνώσης από διαφορετικές πλευρές που συνεργάζονται μεταξύ τους και εμείς να έχουμε ίσως τον συντονισμό ώστε να υπάρξει επιτυχή σχέση εκμάθησης. Τρίτον, θέλουμε να διασφαλίσουμε να υπάρχει καλή γεωγραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων μας και να μην επικεντρωνόμαστε σε ορισμένες χώρες μέλη μόνο, αλλά να καλύπτουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέταρτον, ο ήθιστε, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε περισσότερη πρόσθετη αξία. Έτσι ώστε τα χρήματα τα οποία δίνουμε να αποτελούν πρόσθετη αξία για ολόκληρη την Ευρώπη εκπονώντας τις σωστές ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, και, και αναφέρθηκε στον αντίκτυπο. Όντως, ο αντίκτυπος είναι αυτό στο οποίο θα δώσουμε σημασία. Είναι δύσκολο βέβαια να υπολογίσουμε μέσα σε μια χρονιά τον αντίκτυπο μας στην εκπαίδευση. Χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτόν τον αντίκτυπο. Όμως θέλουμε να πλησιάσουν πιο πολύ οι Ευρωπαίοι την αναπτυξιακή παιδεία και αυτό είναι κάτι που παίρνει χρόνο. Γίνεται σιγά σιγά. Το αποτέλεσμα μέχρι τώρα είναι καλό. Τώρα το να πούμε ότι αυτό έγινε επειδή έχουμε κάνει το ένα ή το άλλο, αυτό είναι βέβαια λίγο δύσκολο. Στην περίοδο κρίσης που βρισκόμαστε, σίγουρα δεν πάμε άσχημα. Θα τελειώσω και με ένα σχόλιο για το περιεχόμενο τώρα. Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της αναπτυξιακής εκπαίδευσης. Όλοι είπαν εδώ ότι δεν πρέπει να πρόκειται μόνο για φιλανθρωπία. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με αυτό. Κάποιο είπε ότι η σχέση ανάμεσα σε αυτόν που ε, έχει την ε, δυνατότητα να δώσει και σε αυτόν που είναι ευγνώμων να πάρει είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει γιατί και οι δύο παίρνουν και οι δύο δίνουν. Το ξέρουμε αυτό και από τις χώρες BRICS και στο κάτω-κάτω και ορισμένοι από αυτού που παίρνουν δεν νιώθουν πια τόση ευγνωμοσύνη όπω νομίζαμε κάποτε. Άρα δεν είναι μια σχέση που βασίζεται στην φιλανθρωπία. Μ' άρεσε ο ορισμός που άκουσα από την κυρία Λίκοβα για την ευθύνη που έχουμε όλοι μας. Και όντως η παγκόσμια εκπαίδευση είναι ακριβώ αυτό, πως όλοι θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ώστε όλοι σε αυτόν τον κόσμο να ζουν με εξωπρέπεια. Και αυτό πρέπει να περάσουμε στους ε, νέους. Ότι κοιτάξτε, εντάξει, κάναμε κάποια λάθη, ο κόσμος είναι σε όποια χάλια πιστεύουμε ότι βρίσκεται, ε, λοιπόν, εσείς τώρα έχετε τα μέσα για να το διορθώσετε. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει. Ότι δίνουμε στους νέους τα μέσα, τις λύσεις για να φτιάξουν αυτό τον κόσμο. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα, είτε πρόκειται για καταναλωτές, είτε πρόκειται για τουρίστες, είτε πρόκειται για μαθητές, για ενήλικες, για επιχειρηματίες, στον ιδιωτικό τομέα, σε οτιδήποτε και ανασχολείται κανείς με οτιδήποτε και ανασχολείται, είμαστε σε ένα παγκοσμιωμένο κόσμο που σημαίνει ότι ο καθένας έχει τη δικιά του ευθύνη σε αυτόν τον κόσμο για την ανάπτυξη. Και αυτή είναι και η βάση της στρατηγικής μας που θα παρουσιάσει και σύντομα ο κύριος Πίλβαξ και αυτό θα είναι το περιεχόμενο. Ολοκληρώνω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που οργανώσατε την σημαντική αυτή ακρόαση. Άκουσα προσεκτικά όλους σας. Και να ξέρετε πώς θα αναλάβουμε πολλές δραστηριότητες πάνω σε αυτό το τομέα μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σμιτ για τις παρατηρήσεις για την Επιτροπή. Τώρα το λόγο έχουν οι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Καλύτερο ήταν να συγκεντρώσουμε όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ε, για όλους ε, τους ε, ομιλητές και να έχουμε απαντήσει στο τέλος. Κύριε Σκάλα, πρώτα, πρώτα. Ευχαριστώ. Πολλοί από τους εκπροσώπους αναφέραν τι έκαναν στην πατρίδα τους, τι έκαναν σε εθνικό επίπεδο. Πολύ καλά όλα αυτά και όλοι αναφερθήκατε στη μέθοδο της ε, αναθεώρησης βάσει ισοτήμων, του peer review. Αυτό το peer review τι έδειξε. Τι είδατε ότι ας πούμε πάει καλά από εδώ, αυτό μας κατέγει, εκείνο μας κατέκριναν τα άλλα Τι συμπεράσματα συνάγεται δηλαδή από αυτό το peer review και τι κάνατε για αυτά τα συμπεράσματα. Αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Συμφωνώ πολύ με την πρόταση να υπάρξει μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική και συντονισμός. Αλλά το ερώτημα που πάντα ανακύπτει είναι τα κράτη-μέλη τι λένε. Είναι καλή ιδέα. Θέλετε να σας συντονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ερώτημα και προς την Επιτροπή. Είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε και να υλοποιήσετε, μια, να υλοποιήσετε μια κοινή στρατηγική που θα ήταν δεσμευτική, όχι μόνο ωραίες ασκήσεις επί χάρτου χωρίς ουσιαστική δράση που δεν βοηθάνε. Και προς την Επιτροπή μια ερώτηση. Ακούσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πολιετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα το λάβετε υπόψη, υπόψη σας όταν παρουσιάσετε το σχετικό κείμενο. Τι, πρόταση, τι έχετε κάνει σχετικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Λουβίν και μετά ο κύριος Γκέρντ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος έθεσε τα πιο σημαντικά ερωτήματα και με την ίδια ευκαιρία θέλω να επαναλάβω την ερώτηση που είχα θέσει και στην προηγούμενη, στο προηγούμενο πάνελ για το περιεχόμενο της ε, αναπτυξιακής εκπαίδευσης. Όταν φτάνουμε στο επίπεδο ανάληψης δράσης, όχι σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε κρατικό επίπεδο. Και γνωρίζοντας ότι προχωρούμε προς μια παγκόσμια κοινωνία και ότι θέλουμε να προωθήσουμε αυτή την παγκόσμια εικόνα του πολίτη, υπάρχει προφανής έλλειψη θεσμών με, με ουσιαστικές αρμοδιότητες. Υπάρχει ο ΙΕ, υπάρχουν οι οι υπηρεσίες περιβάλλοντος κλπ. Αλλά έχουμε ανησυχητικά μηνύματα κενών σε συγκεκριμένες ε, κυβερνήσεις. Δείτε τι γίνεται στη Σομαλία, δείτε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο με περιοχές που δεν, ε, διεθνών υδάτων που δεν έχουν καμία διακυβέρνηση. Αυτά τα ζητήματα θα τεθούν ενώ από τις επόμενες γενιές. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική παράμετρο της αναπτυξιακής εκπαίδευσης για τις επόμενες γενναίες. Το είπε και η Επιτροπή βέβαια. Δεν μπορούμε να τους πούμε κοιτάξτε τα κάναμε θάλασσα, φτιάξτε τα εσείς σε ατομικό επίπεδο. Μπορεί να το πούμε σε ατομικό, αλλά σε θεσμικό επίπεδο τι μπορούμε να προσφέρουμε θεσμικά, δηλαδή κάποια όργανα, κάποιους θεσμούς που μπορούσαν να διορθώσουν το χάος που δημιουργήσαμε. κύριος Γκέρεντ. Ευχαριστώ. Είναι τεράστιο το θέμα και θα προσπαθήσω να το περιγράψω με τρία σημεία. Πρώτον, ενιολογικά, προσεκτικά. Αναπτυξιακή εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι συνώνυμο δογματικής, ε, δογματικής παιδείας. Δεν πρέπει να δημιουργούμε δομές που δεν θα μπορούν να αλλάξουν, αλλά πρέπει να περιλάβουμε, να ορίσουμε το περιεχόμενο. Εάν γίνει δεκτή η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Αναπτυξιακή Παιδεία από την Κοινωνία των Πολιτών, τόσο το καλύτερο. Πιστεύω ότι υπάρχουν μέτρα που θα επιτρέπουν να έρθουν πιο κοντά οι απόψεις. ο διαρθρωμένος διάλογος στον οποίο μετήχαμε ως εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου η κυρία Κέλλα και εγώ και άλλωστε στη Βουδαπέστη ο Επίτροπος κ. Σπίμπαλξ είχε αναγγείλει την έκδοση μιας ανακοίνωσης για τη συνέχεια της, ε, του εγχειρήματο αυτού που είναι πολύ εύλογο. Δεύτερο, χρηματοδότηση. Καλές οι ιδέες αλλά χρειαζόμαστε και λάδι στον κινητήρα. Στην ευρωπαϊκή λοιπόν στρατηγική μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εμένα, με, με, εγώ απεχθάνομαι τις μεγάλες στρατηγικές. Όταν δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε λέμε στρατηγική. Χρηματοδοτούμε μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης ή μέσω του προϋπολογισμού των κρατών μελών ή μέσω και των δύο. Κάπως και κάποιος πρέπει να συμφωνήσει για την προστιθέμενη αξία που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρηματοδοτήσει ή να συγχρηματοδοτήσει το κέντρο ε, του που το θεωρεί διότι ε, μπορεί να λειτουργήσει καλά. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να κρατήσουν ένα ποσοστό χ με στόχο την ευαισθητοποίηση που είναι ο κύριος στόχος της ε, εκπαίδευσης για την ανάπτυξη. Να επιτρέψει δηλαδή στους φορείς να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη της Ευρώπης και να δημιουργήσουν και κάποια πολιτικά κίνητα. Τρίτο θέμα και είναι σημαντικό αν και επειδή θα καθυστερημένο δεν ξέρω αν το είδατε ήδη. Υπάρχουν και εταίροι στο Νότο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια στρατηγική, η στρατηγική πρέπει να στηρίζεται σε μια σειρά κοιώνων που περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ε, στη σύμβαση του Κοτονού και που προβλέπει την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών ως έναν από τους νέους παράγοντες στον τομέα της ανάπτυξης. Η κοινωνία των πολιτών στις χώρες ΑΚΕ εννοώ. Και χρειαζόμαστε πραγματικά, εάν θέλουμε να προωθήσουμε ε, να προχωρήσουμε οικονομικά θα πρέπει στις δικαιούχους χώρες να υπάρχει μια κοινωνία των πολιτών που θα είναι ικανή να καλύψει τις ανεπάρκειες σε θέματα διακυβέρνησης του κράτους. Πρέπει να υπάρχει ένα κριτικό αντίβαρο που είτε θα που, συχνά είτε παραμερίζεται είτε απορρίπτεται ρητά από τις κυβερνήσεις. Η στρατηγική λοιπόν πρέπει στον τομέα της εταιρικής σχέσης με τις χώρες του Νότου θα πρέπει να στοχεύει εκεί, να προχωρήσει σε έναν κάποιο απολογισμό της ε, συνεργασίας μεταξύ χωρών ΑΚΕ και Ένωσης. Τι έγινε στον τομέα τη οικοδόμησης τη χώρα ΑΚΕ τη κοινωνία κοινωνία των πολιτών. Έχω μια ασαφή εικόνα που δεν είναι καθησυχαστική κατά βάση. Αυτό το ζήτημα νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πρώτο. Ούτως ώστε οι ανεπάρκειε αυτές, και είμαι βέβαιος ότι οι ανεπάρκειε αυτέ υφίστανται, να συμπεριληφθούν στις συζητήσεις μας, ούτως ώστε να διαγνώσουμε τις αδυναμίες και να τις θεραπεύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Γκέρεντ. Πέντε ομιλητές έχουμε τώρα, ήθελα να απαντήσει και η Επιτροπή. Θέλετε? Τρία λεπτά ο καθένας λοιπόν από τους πέντε ομιλητές. Κύριε Σμιτ. Πρώτα οι πυρογνώμονε. Ανάποδα. Πρώτα Λαπαλάιεν. Um, Να απαντήσω στο θέμα της ευθύνης. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το ρόλο του κράτους. Αλλά ποιο είναι κράτο. Κράτο είναι οι πολίτε. Άρα ο κάθε άνθρωπο πρέπει να ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο μέχρι επάνω τι κρατικέ δομέ. Εγώ έτσι βλέπω την στρατηγική μας για την εμπλοκή των διαφόρων ε, δομών και δυνατοτήτων. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι και η Ένωση χρειάζεται για να έχει μια αναπτυξιακή, μια στρατηγική αναπτυξιακή εκπαίδευση. Υπάρχουν όντω πολλές συμφωνίες. Αλλά τι χρειαζόμαστε κυρίως, χρειαζόμαστε ένα πολιτικά δεσμευτικό σύστημα που θα πάρει τα πολλά παραδείγματα που υπάρχουν και θα τα ενσωματώσει σε ένα ενιαίο πακέτο. Προφανώς υπάρχει συμπληρωματικότητα των κρατών μελών. Προφανώς χρειάζεται να λειτουργήσει η καλύτερη κοινωνία των πολιτών. Αλλά αυτό το παιχνίδι το κάνουμε 10-20 χρόνια. Πρέπει να σταματήσουμε την πολλαπλότητα, να βάλουμε όλες τις δραστηριότητες μας σε ένα πακέτο και με αυτό το πακέτο να δουλέψουμε. Συμφωνία Κοτονού. Όντως είναι πολύ σημαντική. Εκεί χρειάζεται μια παγκόσμια κοινωνία των πολιτών. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για μας δεν είναι μόνο οι κοινωνίε των πολιτών, αλλά είναι τα κράτη, είναι οι κοινωνίε των πολιτών και είναι οι ίδιοι οι πολίτε. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε την κοινωνία των πολιτών, ούτε μπορούμε να απομονώσουμε τη στρατηγική της Ένωση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριο Σκούμπερ. Ναι, Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί, μια νέα στρατηγική και ε, υπάρχει και η εξέταση από τους ομολόγους μας. Εγώ σύμφωνο ότι χρειάζονται προφανώς η Ευρώπη να συνεργάζεται, να υπάρχει συνεργασία δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συντονισμός με ό,τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και μιλώ όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για το Συμβούλιο της Ευρώπης και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διότι έτσι μπορούμε να προωθούμε τα θέματα που εξετάσσονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης και να τα επαναφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα στρέφομαι και συνεχίζω στα γαλλικά που είναι η μητρική μου γλώσσα για να την προωθήσω εφόσον είναι σημαντική η γλώσσα και υπάρχουν δύο βασικά θέματα η χρηματοδότηση διότι κανόνες δεν μπορεί να παραβλέψει ε, την ε, χρηματοοικονομική κρίση στα κράτη-μέλη και τα κράτη της Ευρώπης και του Βορρά και του Νότου ε, πρέπει να υποστούν όλες τις επιπτώσεις και γι' αυτό πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα από την άποψή μας. Η σημασία της ε, κοινωνία των πολιτών επίσης είναι ουσιαστική διότι έχουν γίνει προσπάθειες μέσω ενός ο προγράμματος που αναφέρεται στην Ευρωαφρικανική Νεολαία προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τις οργανώσεις νεολαία στην Αφρική βάσει των προτύπων που ισχύουν στην Ευρώπη και όλα αυτά έχουν γίνει με, με συντονισμό αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα όταν πρόκειται για χώρες οι οποίες δεν είναι δημοκρατικές γιατί δεν μπορούμε να βρούμε οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που να είναι ανεξάρτητες από την εξουσία αλλά υπάρχει μία μεταστροφή και η δημιουργία μιας μεγάλης κοινωνίας των πολιτών μπορεί να γίνει στη μετάβαση αυτή προς τη δημοκρατία η οποία διεξάγεται σε πολλές χώρες. Ευχαριστώ κύριε Χούμπερ. Ο κύριος Χαρτμάγερ. Εμένα τα γαλλικά μου είναι πολύ φτωχά, οπότε θα συνεχίσω αγγλικά που δεν είναι η μητρική μου, σχετικά με την αξιολόγηση από τους ομοτήμους peer review. Ε, έχουμε διάφορες εμπειρίες σε διάφορες χώρες αλλά υπάρχει μία έλλειψη συνεκτικότητος ε, διότι στον τομέα των αναπτυξιακό και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνεκτικότητα και αυτό ισχύει σε διάφορα θέματα. Υπάρχει μία έλλειψη συντονισμού. Δεν είμαστε παντού τυχεροί όπως στην Πολωνία όπου ο Υπουργός Παιδείας και Υπουργός Εξωτερικών έχουν τα γραφεία τους σε διπλανά κτίρια αλλά σε πολλές χώρες οι υπηρεσίες δεν συνομιλούν, δεν συντονίζονται, δεν υπάρχουν ε, χρήματα, δεν είναι όλοι στην ευτυχή ε, θέση της Σκανδιναβίας και της Ολλανδίας όπου υπάρχει ευρεία χρηματοδότηση για τον τομέα αυτό σε πολλά μέρη υπάρχει έλλειψη ε, πόρων χρειάζεται λοιπόν περισσότερο συντονισμός και αυτό είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτό. Ε, όσον αφορά το περιεχόμενο της παιδείας νομίζω ότι υπάρχει μία τάση δηλαδή να τονίζουμε υπερβολικά την ε, εκπαίδευση των ατόμων και υπάρχουν δομικές αλλαγές για δομικά στοιχεία τα οποία παραβλέπονται και αυτό είναι μία τάση η οποία ε, αναφέρεται σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή οι υπεύθυνοι ε, είναι ε, μεν ε, μία ε, κοινή προσπάθεια αλλά δεν μπορούν ε, μόνο αυτοί να λύσουν τα δομικά προβλήματα που υπάρχουν και οι δομές δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν την έλλειψη πολιτικής. Δεν μπορεί η παιδεία να φέρει την ευθύνη των αλλαγών. Μπορεί να να προωθήσει τις αλλαγές, να προωθήσει δεξιότητες ε, και γνώσεις που θα επιτρέψουν ε, εις ε, τα άτομα να συμμετάσχουν στις αλλαγές αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλα θέματα και δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες της κοινωνίας των πολιτών είναι ένα υπερβολικό φορτίο το οποίο δεν μπορεί να αναλάβει. Ευχαριστώ κύριε Χαρτμάιερ και τέλος ο κύριος Στανό τη της Πολωνίας όπου είναι τυχερό στα γραφεία του, ε, της παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών να είναι δίπλα-δίπλα. Πιστεύω και εγώ εις, ε, την ε, συνολική παιδεία η οποία θα έχει σχέση με την ε, ευρωπαϊκή με τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα πρέπει όμως καταρχήν να καταρτήσουμε μία κοινή δεσμευτική στρατηγική. Επαναλαμβάνω λοιπόν και πάλι ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για δεσμετικές ε, στρατηγικές όπως ε, το κάνουμε για τα μαθηματικά. Πρέπει λοιπόν η ε, εκπαίδευση του πολίτη να γίνει αλλά είναι ένα λεπτό θέμα. Συζητάμε με τους Γερμανούς γειτόνους μας πώς μπορούμε να έχουμε ένα κοινό βιβλίο Μουσείο Ιστορίας κοινό μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας για να γνωρίζουμε ο καθένας πώς σκέφτεται η γειτονική μας χώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για την παιδεία σε μια κατάσταση όπου τα συστήματά μας τα εκπαιδευτικά είναι τελείως διαφορετικά. Ο ρόλος του γονιού, της ε, ε, τοπικής κοινωνίας, της κυβερνίας, στα στα διάφορα κράτη-μέλη είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση είναι μια καλή άσκηση και πιστεύω ότι όλοι όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ετοιμαστούν να εξελίξουν καλύτερα την κατάσταση διότι αυτή τη στιγμή δεν προχωρούμε σωστά. Το δεύτερο βασικό στοιχείο, εάν θέλουμε να αναπτύξουμε κάτι το οποίο είναι ε, κοινό, χρειαζόμαστε ομολόγους και από τον Νότο, αλλά καλά και από την κοινωνία των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδίως από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στην πραγματική ε, δράση εις ε, τον Νότο ε, στα πλαίσια της συνεργασίας. Δεν συμμεριζόμαστε όλοι τα έγγραφά μας, αλλά καταρχήν πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται επί τόπου και τέλος χρειαζόμαστε μια βασική ε, ε, ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσουμε δηλαδή να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να προχωρήσουμε αλλά είμαστε ε, βέβαιοι ότι ε, η κοινωνία η σχολική θα κάνει κάτι για τους ομολόγους ε, στην Αφρική ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα συμβάλλει στην συνεργασία με κάποια κάποια περιοχή στο ε, νότιο ειρηνικό. Αν αυτό μπορέσει να γίνει τότε όντως η συνεργασία θα είναι θετική και επικοδομητική. Και Πρέπει να σας πω ότι είμαι βέβαιος ότι αν η παιδεία παραμείνει στην κορυφή της ημερησίας διατάξεως θα μπορέσει να προωθήσει και την αναπτυξιακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ κύριε Στανόφσκι. Σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ μερικά σχόλια αλλά πρώτα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, ε, είναι υποχρέωση να παρέμβω αλλά καταρχήν θα υπάρξει μία ε, επαφή με τις τοπικές αρχές την οποία έχουμε υποσχεθεί και στον τομέα αυτό θα προωθήσουμε την αναπτυξιακή παιδεία. Πιστεύω ότι στο θέμα αυτό υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση και το βασικό είναι να ξεκινήσουμε την εφαρμογή των συστάσεων στις οποίες κατέληξε η μελέτη. Επ' αυτού έχω ακούσει πολλά καλά νέα τα οποία θέλω να προωθήσω. Θέλω συγχρόνως να ε, συμφωνήσω για το διάγραμμα της στρατηγικής η οποία επαναλαμβάνει πολλά πράγματα οποία και εμείς προωθούμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κινηθούμε όλοι από κοινού και τέλος θα αφήσω το θέμα αυτό ή στους ε, επικεφαλείς ε, ε, των διαφόρων τομέων διότι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν. Χρειάζεται μία στρατηγική προσέγγιση και τέλος η ερώτηση ήταν τι θα συμπεριληφθεί στο πολυετές πρόγραμμα και ε, όπως σας είπα θα υπάρξει ένα πρόγραμμα το Δεκέμβριο αλλά τελικώς το θέμα αυτό θα έχει δύο πτυχές καταρχήν ε, για τα ε, συνολικά δημόσια αγαθά και δεύτερον ε, τοπική αυτοδιοίκηση και μη κρατικοί παράγοντες όπου θα υπάρξει μία αύξηση 20% για να μπορέσουμε να προωθήσουμε καλύτερα την αναπτυξιακή παιδεία. Πιστεύω όμως και θα συμφωνήσετε ότι επειδή αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, για το mainstreaming, για ε, τα προγράμματα τα εθνικά της ε, εκπαίδευσης, παρόλο που προσφέρουμε μία αύξηση ε, ε, του, κατά 15-20% δεν θα επαρκέσει. Και έρχομαι τώρα στο σχολικό πρόγραμμα. Ε, πάντοτε ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσουμε, αλλά αν δεν υπάρχει η θετική πρόθεση από τους ομολόγους, ε, δεν θα μπορέσουμε να το, ε, να το προωθήσουμε και ε, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί για το πόσο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα, θα απευθυνθώ όμως στο Γενικό Διευθυντή για πολιτισμό και εκπαίδευση για να επανέλθω και να σας πω πώς πόσο ρεαλιστικά θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη ε, να ε, ε, να συμβάλλουν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να ακούσουμε την Επιτροπή και τώρα είναι βασικό και ε, εφόσον υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή μπορώ να προχωρήσω στις παρατηρήσεις μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε εδώ σήμερα και συζητήσαμε διάφορες εμπειρίες και παραδείγματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της συνεργασίας. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η εκπαίδευση για την ανάπτυξη αποτελεί στοιχείο κλειδί προκειμένου να ε, χτίσουμε την ε, συνειδητοποίηση, την εγρήγορση που χρειάζεται στον κόσμο υπέρ της ανάπτυξης. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, εκπαίδευση της ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να λάβει, να αναλάβει μάλλον τις ευθύνες του και να αναλάβει και την ίδια του την ανάπτυξη, ιδίως στις υπανάπτυξη χώρες. Και αυτό θα γίνει μέσω ε, δέσμευσης από της διεθνούς κοινότητας. Χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πολιτική δράση και δέσμευση οικονομική προκειμένου να πετύχουμε περισσότερα για την ανάπτυξη στη νέα περίοδο. Είμαι σίγουρος ότι η ακρόαση αυτή συνεισέφερε θετικά στη συζήτηση για τις μελλοντικέ προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να σας πω ότι θα μελετήσουμε σοβαρά τη δυνατότητα να αφιερώσουμε μια έκθεση στην ε, εκπαίδευση για την ανάπτυξη σύντομα ώστε να βοηθήσουμε και εμείς την εκπόνηση μελλοντικών ε, ευρωπαϊκών πολιτικών υπέρ της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη, υπέρ της σχετικής μας στρατηγικής και υπέρ περισσότερων οικονομικών μέσων για την ανάπτυξη. Εφόσον όλες οι πλευρές ε, σταθούν στην ίδια πλευρά, θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά. Θέλω να ολοκληρώσω θυμίζοντας τι είπε ο Παύλο Φορέρο, ο οποίος είπε ότι η εκπαίδευση ή που λειτουργεί σαν ένα εργαλείο, σαν ένα μέσο που χρησιμεύει για να διευκολύνουμε την ανάπτυξη της μελλοντική ε, γενιάς, αποφεύγοντας το status quo, ή θα αποτελέσει την πρακτική για την ελευθερία βάσει της οποίας άντρες και γυναίκες με δημιουργικότητα και φαντασία θα διαπιστώσουν πώς μπορούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία του ίδιου τους του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσοι πήρατε μέρος στην ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ και τους Δερμηνείς, λέει ο μιλητής. Και ευχαριστώ και τον συμπρόεδρό μου εδώ.